Uh, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, θα ήθελα να κήξω την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης και να σας καλωσορίσω όλες και όλους. Τρέχει ο χρόνος. Θα θυμάστε κύριε Επίτροπε, όταν είχατε έλθει πριν από ένα χρόνο εδώ μας παρουσιάσετε την νομοθετική δεσμέτρων και τώρα είμαστε μέσω διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Έχουμε τακτικές συναντήσεις και ελπίζω σε κάποιους μήνες, μακάρι να μπορούσα να πω στο τέλος του χρόνου, αλλά καλό θα ήταν να μην κάνουμε τέτοιες δεσμεύσεις, όπως μου είπατε και εσείς, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις για τα νομοθετικά ζητήματα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πάντως Για πρώτη φορά ίσως ξέρετε ότι ως ευρωβουλευτές είμαστε συνομοθέτες πλήρως. Άρα είμαστε σε ισότιμη θέση με το Συμβούλιο. Γιατί πλέον η κανονική νομοθετική διαδικασία ισχύει και για την ε, νομοθετική δεσμή μέτρων. Θα ήθελα να σας πω ότι στο νομοθετικό πλαίσιο στηρίζουμε πλήρως την Κομισιόν σε πολλά σημεία. Επίσης, για πολλά ζητήματα έχουμε ευθυγραμμιστεί και με το Συμβούλιο, αλλά υπάρχουν παρόλα αυτά ορισμένα σημαντικά στοιχεία για το μελλοντικό πλαίσιο, τη μελλοντική πολιτική, επί των οποίων ακόμη εργαζόμαστε για να βρούμε μια καλή συμμεβαστική λύση. Πρέπει να σας πω ότι στηρίζουμε όλοι στεναρά τη νέα προσέγγιση την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήτι έναν γενικό κανονισμό ομπρέλα που θα καλύπτει όλα τα ταμεία, ώστε να εξασφαλιστεί συνεκτικότητα, συνέπεια μεταξύ των κανόνων που ισχύουν για τα ταμεία, αλλά και συνέργειες ε, για την χρήση των ε, ταμείων ως εκπλήρωση των βασικών στόχων του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης, στηρίζουμε την ιδέα ένα νέο έγγραφο να αντικαταστήσει ε, τα εθνικά ΕΣΠΑ και να έχουμε ένα ε, κοινό στρατηγικό πλαίσιο που θα καλύπτει όλα τα ταμεία. Και έτσι θα έχουμε κάποιες οριζόντιες αρχές για τα ταμεία και θα έχουμε και ένα καλό θεμέλιο, μια καλή βάση για καλύτερο συντονισμό μεταξύ της πολιτικής συνοχής και άλλων χρηματοοικονομικών μέσων που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη. Ενώ και τη στρατηγική του 2020, αλλά και κάποια άλλα στοιχεία, κάποια ε, μηχανισμούς όπως είναι το Connecting Europe, ε, συνδέοντας την Ευρώπη δηλαδή, ή κάποια άλλα ε, στοιχεία που έχουν να κάνουν με τα κοινωνικά θέματα, τι κοινωνικέ αλλαγές και πρέπει να σας πω ότι είμαστε πρωταθλητές εδώ ε, στις ενισχυμένε εταιρικέ σχέσεις ε, και συνεργασίες όπως προτείνεται σε αυτό το νέο πλαίσιο πολιτική. Ελπίζουμε όλα τα σημαντικά ζητήματα και για τον προγραμματισμό και για την υλοποίηση να συναποφασίζονται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και να υπάρχει ισχυρή συμμετοχή των τοπικών περιφερειακών αρχών και άλλων εταίρων που θέλουμε να προσδιορίζονται ακριβώς και στον κανονισμό ώστε να έχουμε και εταιρική σχέση με τις διάφορες οργανώσεις εκπροσώπους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Ελπίζουμε όλοι αυτοί να μπορέσουν να λάβουν μέρος στην εταιρική αυτή σχέση και στις σχετικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Θέλουμε λοιπόν να ενισχυθεί η εταιρική σχέση σε αυτό το νέο πλαίσιο πολιτικής. Στηρίζουμε επίσης και την εδαφική διάσταση της πολιτικής. Στόχος μας στις διαπραγματεύσεις είναι να δοθεί ένας ισχυρότερος ρόλος στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και αρχές. Αυτό ελπίζουμε να γίνει πράξη. Ελπίζουμε επίσης η εδαφική διάσταση όπως παρουσιάζεται με τα νέα μέσα που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη, κινητοποίηση τοπική ανάπτυξη. Έχουμε μια πρόταση τη Κομισιόν, περιλαμβάνει 7 νέα μέσα τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική διάσταση της ανάπτυξη, των τρελατικών αλλαγών, με ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των εταίρων. Αυτό είναι ένα νέο χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό της πολιτικής αυτής. Στηρίζουμε επίσης και την ανάγκη συγκέντρωση της χρηματοδότησης. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο βέβαια. Και από την εμπειρία μας μέχρι τώρα, από την πολιτική αυτή, χρειάζεται διαφοροποίηση. Αλλά για να βγούμε από την κρίση θα χρειαστούν πολλές δράσεις στοχευμένες ακριβώς στις τοπικές περιφερειακές ιδιαιτερότητες ε, και σε αστικό επίπεδο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στηρίζουμε λοιπόν τη συγκέντρωση ταυτόχρονα όμως με τις προτάσεις μας και με την εντολή μας προσπαθούμε να δώσουμε και μεγαλύτερη ευελιξία στη διάσταση αυτή της πολιτικής, διότι πιστεύουμε ότι οι περιφέρειες, οι δήμοι πρέπει να έχουν περισσότερη ελευθερία για να μπορούν να προσαρμόζουν την πολιτική στα, στις ιδιαιτερότητες, στα χαρακτηριστικά τους και να αξιοποιούν καλύτερα το δυναμικό τους για μεγαλύτερη ανάπτυξη και βιώσιμη απασχόληση. Και άλλωστε με την κρίση πλήττονται με κάπως ιδιαίτερο θα έλεγα τρόπο οι διάφορες περιφέρειες. Πρέπει να είμαστε λοιπόν εδαφικά πιο ευαίσθητοι. Άλλος στόχος είναι η ενισχυμένη συνεργασία για να δώσουμε όθηση σε μια θετική αλλαγή στην ανάπτυξη περισσότερες θέσεις εργασίας. Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη σύγκληση και γι' αυτό θέλουμε και το μηχανισμό σύγκλησης στην Ευρώπη να τον ενισχύσουμε, γιατί βλέπουμε μια επιβράδυνση ξεκάθαρη τα τελευταία δέκα χρόνια. Βέβαια πρέπει να πω ότι ακόμη και το καλύτερο δυνατό πλαίσιο που από κοινού θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με την συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και των εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τι έχουμε στενή συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, να σας ενημερώσω. Ακόμα λοιπόν και αν καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό πλαίσιο, και πάντα θα πρέπει το επόμενο πλαίσιο να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση αυτή η αρχή. Παρόλα αυτά, θα τα καταφέρουμε μόνο αν έχουμε και έναν αξιοπρεπή προπολογισμό για τα επόμενα έτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο-τρία ζητήματα σχετικά θα ήθελα να αναφέρω, γιατί θέλω να σας πείσω ότι Head of us of budget consolidation at national... σίγουρα χρειάζεται να γίνει δημοσιονομική προσαρμογή. Για να γίνει αυτό θα πρέπει το, βιο... το χρέος να καταστεί βιώσιμο, να γίνουν ε, οικονομίες. Παρά τη λογική αυτή όμως εγώ νομίζω ότι πρέπει να στοχεύσουμε προς έναν ευρωπαϊκό προϋπολισμό που πραγματικά να μπορεί να παράγει θέσεις εργασίας. Και σίγουρα χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα χρηματοδότηση, αυτό το γνωρίζουν οι ειδικοί και πρέπει να καταλάβουμε ότι επειδή γίνεται αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή και εξυγίανση σε εθνικό επίπεδο, εδώ δεν πρέπει να έχουμε την ίδια ακριβώς λογική, γιατί καταλήτης για επενδύσεις στην Ευρώπη είναι οι πόροι, τα δημόσιοι πόροι και ο Ευρωπαϊκό προλογισμός πρέπει να έχει την υπόψη είναι προσανατολισμένος σε επενδύσεις, επενδυτικός προϋπολογισμός. Μόνο το 5% λίγο πολύ του προϋπολογισμού πραγματικά πηγαίνει ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες. Ο περισσότερος προπολογισμός, το 95% είναι επενδύσεις ε, στις πόλεις, ε, στην περιφέρεια, στα κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, γιατί υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα. τα οποία προβάλλονται και από τα ΜΜΕ. Να πω κάτι ακόμη. Αυτή όλη η διαδικασία της νοσομικής εξυγίασης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα έχει και εκεί επιπτώσεις. Χρειάζεται συγχρηματοδότηση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ήδη σήμερα βλέπουμε ότι και ε, τα θέματα δημοσιονομικής ευθύνης και λογοδοσίας έχουν το ρόλο τους. Υπάρχουν προκλήσεις και σε αυτό το πεδίο. Τοπικοί, περιφερειακοί προϋπολογισμοί συρρυκνούνται. Και εκεί θα υπάρξει πρόβλημα με τη συγχρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο. Άρα διαγράφεται και μία απειλή οι ευρωπαϊκές επενδύσεις να μην είναι σε θέση να γίνουν πράξη. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα και στο επίπεδο των Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει να σκεφτούμε αυτή την πρόκληση πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Το τελευταίο μήνυμα που θέλω να σας δώσω, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, είναι ότι είμαστε στην ε, διαδικασία της ε, διαπραγμάτευσης για τον περιπολισμό του 2013 και για την τροποποίηση του τρέχοντος προπολογισμού. Ίσως ο Επίτροπος, δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί να είναι όσο ανοιχτός ε, όσο είμαι εγώ, αλλά και να σας τα πει όλα ειλικρινά, αλλά θέλουμε σε ό,τι αφορά τα ήδη σε εξέλιξη έργα να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ που μπορεί να μπλοκαριστούν. Επειδή έχουμε πάρα πολύ μικρό προϋπολογισμό και το 2012. Άρα έχουμε και αυτή την πρόκληση να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε τον τρέχοντα προϋπολογισμό για να χρηματοδοτήσουμε project τα οποία θα μπορούσαν να, ίσως να διακοπούν, να ανασταλούν ή τέλος πάντων έχουν μπλοκαριστεί. Είναι σημαντικό να έχουμε αυτό το διορθωτικό προπολογισμό, γιατί οι πολιτικέ πρέπει να φέρουν αποτελέσματα. Χωρί χρήματα, χωρί χρηματοδότηση δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη απασχόληση και περισσότερη ανάπτυξη. Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνω την εισαγωγική μου παρέμβαση και θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα τον Επίτροπο, τον αρμόδιο για την περιφερειακή πολιτική, τον κύριο Γιωάννη Χάν, να μας μιλήσει, να μας μεταφέρει τις δικές του ιδέες. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ, Ντανούτα, και καλημέρα και από πλευρά μου. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους εδώ παρόντες, ιδιαίτερα τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι η τέταρτη φορά που έχουμε αυτή την διακοινοβουλευτική συνεδρίαση και έτσι έχω και εγώ την ευκαιρία να συζητήσω θέματα της ε, περιφερειακής πολιτικής μαζί σας. Είχαμε και τις ε, Open Days, ανοιχτές ημέρες εδώ στις Βρυξέλλες, με μια σειρά από σεμινάρια, εκδηλώσεις. Ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με δραστηριότητες. Η προκάτοχος και τωρινή πρόεδρος Επιτροπής των Περιφερειακών Θεμάτων, κυρία Αντωνούτα Χούμπνερ, ήδη περιέγραψε την κατάσταση σχετική με την περιφερειακή πολιτική και όσο και αν είναι ασύνηθες. Πρέπει να ομολογήσω ότι μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε μια ταύτιση απόψεων και προτάσεις κοινέ για, την, ε, για τις εξελίξεις στην περιφερειακή πολιτική και ιδιαίτερος το θέμα της χρηματοδότησης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το να μπορώ να έχω μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας ο πρόεδρος Φαν Ρόμποϊ έχει προβλέψει σε ένα ειδικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 21-22 ε, Νοεμβρίου ε, την συζήτηση των θεμάτων αυτών ιδιαίτερα και νομίζω ότι πρόκειται για μια απόφαση να προχωρήσουμε, σηματοδοτείται έτσι μια απόφαση να προχωρήσουμε μέχρι το χρόνο. της πρωτεύουσας, της πρωτεύουσας των κρατών μελών ε, πρέπει να κάνουμε προσπάθειες προκειμένου να υποβοηθήσουμε και την περιφερειακή πολιτική ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Και γι' αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι κάθε επαφή που έχουμε εδώ στις Βρυξέλλες φυσικά αλλά εν γέννη ε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και γι' αυτό πάντοτε αισθανόμαστε μεγάλη χαρά για να συζητούμε και για να αντιμετωπίσουμε κάποιες τάσεις που θα μπορούσα να εντοπίσω για περικοπές στον τομέα αυτών. Και ξεκινώντας θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ κεντρική σημασία θέμα. Ζητήματα τα οποία έχουν νομίζω διαμορφώσει κατά κάποιο τρόπο την συζήτηση. Το πλαίσιο αναφοράς για τα δεύτερη ταμεία, τις ε, εταιρικές σχέσεις και το πρόβλημα της ε, περικοπής στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, στον προϋπολογισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διαπραγματεύσει λοιπόν για το νομικό πλαίσιο για την προσεχή πολιτικής συνοχής έχουν προχωρήσει κατά την ε, εκτίμησή μου αρκετά ικανοποιητικά και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως η έκθεση με την οποία προσδιορίστηκε η δυνατότητα της εξέταση ε, πρώιμη εξέταση των προτάσεων της Ευρωπαϊκή Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη αποτελεί μια πολύ καλή εξέλιξη. Έχουμε ήδη το, στον προγραμματισμό μας της τον τριμερή διάλογο. Άρα η συνεργασία και η επαφή μεταξύ των πλευρών μας, των δύο πλευρών, είναι ήδη αρκετά προωθημένη. Εδώ πάνω απ' όλα Θέλουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε ένα στόχο, έχουμε ένα μεγάλο στόχο και θέλουμε το χειρότερο δυνατό καλά αποτελέσματα, αποφάσει που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να είμαστε σε θέση και κατά τη διάρκεια του 2013 και όσο το δυνατόν πιο σύντομα να ε, προβούμε στις ε, λοιπές διαπραγματεύσεις με τις περιφέρειες, τα κράτη-μέλη, ώστε να είμαστε έτοιμοι και κατά το δυνατόν να διαμορφώσουμε απρόσκοπτα τη μετάβαση στη νέα περίοδο από το 2014. Αυτά λοιπόν προς το συμφέρον της ε, διαμόρφωσης του κατάλληλου, της κατάλληλης πρικοδότησης του προπολογισμού, αλλά και του σωστού περιεχομένου για την περιφερειακή πολιτική. Όπως είπα, έχουμε συνένεση μεταξύ μας, σελίδα τη συνένεση. Θα αναφερθώ όμω ε, στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο, καταρχάς, καταρχάς ε, τα ταμεία. Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανάπτυξη Πέθρου, Ταμείο Συνοχής, Ταμεία για την Ανάπτυξη Αλίας. Είναι προτάσεις, είναι ταμεία τα οποία καταγράφονται και σημειώνονται στο πλαίσιο μιας ε, ευρωπαϊκής ενός ευρωπαϊκού προγραμματισμού, ενός ευρωπαϊκού σχεδιασμού, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι κονδύλια παίρνει ποιο ταμείο. Για να αποφεύγουμε τις επικαλύψεις, αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν τομείς τους οποίους δεν θα καλύπτει ούτε το ένα ούτε το άλλο ταμείο ως προς τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Αυτά λοιπόν είναι οι προτάσεις μας για το στρατηγικό, για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ως προς το περιεχόμενο, ως προς την ουσία προβλήματα δεν υπάρχουν. Ε, το ζητούμενο είναι περισσότερο τυπικά πώς θα χειριστούμε το θέμα αυτό του κοινού στρατηγικού πλαισίου και το πώς θα βοηθήσουμε και τα κράτη αλλά και τις περιφέρειες ιδιαίτερα να αντιδράσουν ταχύτερα για να έχουμε χάρη στην καταξουσιοδότηση πράξη την διευθέτηση των ζητημάτων. Ε, και ελπίζω ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις και αντιρρήσεις ε, η πρόταση που προβάλλεται είναι να έχουμε ένα παράρτημα στον κανονισμό με βάση τον οποίο θα μπορεί να λειτουργεί στην ουσία το σύστημα Υπάρχουν κάποιες βασικές ιδέες πάνω στις οποίες θα στηριζόμαστε ασφαλώς στο πλαίσιο αυτού του στρατηγικού πλαισίου και αναλόγως θα μπορούμε να ακολουθούμε για τις βασικές γραμμές τα ε, προκαθορισμένα, για δε τα λοιπά μπορούμε να έχουμε περισσότερη ευελιξία την οποία μας προσφέρουν ή κατεξουσιοδότηση πράξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μια ε, καλή, μια πρακτική λύση, μια εφικτή λύση, έτσι ώστε ο δικαιούχος, αυτός τον οποίο απευθύνονται τελικά αυτά τα προγράμματα, να είναι σε θέση να επωφεληθεί του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Ο άλλος τομέας είναι η συμβάση εταιρική σχέσης όπου θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα ένα θέμα για τις συμβατικές, για τις συμβάσεις εταιρικής υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς και ιδιαίτερη ε, επιθυμία του Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς της περιφερειακής πολιτικής στην διαπραγμάτευση για τις συμβάσεις αυτές. Έτσι θα είμαστε και βέβαιοι ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη αποδοχή αυτών των συμβάσεων και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και στο ρυθμιστικό επίπεδο έχουμε ένα άρθρο για το multi-level governance όπως ονομάζεται, δηλαδή το, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να μεριμνήσουμε στις διαπραγματεύσεις το τοπικό όσο και το περιφερειακό επίπεδο, αλλά και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή, συμμετοχή στις ε, διαπραγματεύσεις. Προτείνω λοιπόν εάν έχετε κάποιες ε, προτάσεις να τις υποβάλλετε. Θα ήθελα τώρα για το δημοσιονομικό πλαίσιο να επισημάνω ότι η κυρία Χιούμπνερ με έχει καλύψει, δεν έχω πολλά να προσθέσω. Ένα ίσως θα μπορούσα να προσθέσω στην, ε, ε, στο θέμα που με απασχολεί ιδιαίτερα, που θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω. Και ξεκινώ λέγοντας ότι από την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στο παρελθόν έχω και με τον περιφερειακό αλλά και με την κεντρική διοίκηση, κυβέρνηση, ιδιαίτερη, ιδιαίτερη εμπειρία και γι' αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος κατά 95% επανέρχεται στα κράτη-μέλη, είτε πρόκειται για πληρωμές, είτε πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης, είτε πρόκειται για, για ε, ε, προγράμματα ενίσχυσης αναπτυξιακής βοήθειας και μόνο 5% μόνο 5% καλύπτει τα το κόστος, το λειτουργικό κόστος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όλων των θεσμικών οργάνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, Ελεκτικού Συνεδρίου, Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες κτλ. Άρα λοιπόν, αν δείτε αυτό τον λόγο, αυτή την αναλογία, 95% που επανέρχεται στα κράτη-μέλη και 5% που είναι το, κόστος γενικής, ε, το γενικό κόστος λειτουργίας, νομίζω ότι μπορούμε να αναγνωριστούμε ως ο φορέας και η διοικητική αρχή ανά τον κόσμο με το χαμηλό ε, με το χαμηλότερο κόστος, ε, με την πιο οικονομική διαμόρφωση, ε, λειτουργία. Και έτσι θα έλεγα ότι αποτελούμε μια πολύ καλή και γη επένδυσε. Και έτσι περνάω στην λέξη επένδυση, ο, ε, ο προϋπολογισμός με τις επενδύσεις, θα επενδύσει στι περιφέρειε, θα επενδύσει στους ανθρώπου, στις δεξιότητες του, στην ανταγωνιστικότητα, στη βελτίωση των δυνατοτήτων ε, τόσο μέσα σε ε, ενδοευρωπαϊκό επίπεδο και ισορροπίε όσο και ανά τον κόσμο. Εάν αναλογιστούμε ότι έχουμε πέντε 500 εκατομμύρια πολίτες εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκπροσωπούμε μόνο 7% του παγκόσμιου πληθυσμού και όμως αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας παράγων στη διεθνή σκηνή με μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 1 τέταρτο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και νομίζω ότι μπορούμε όχι μόνο είμαστε περήφανοι για την παρουσία μας αυτή ε, στη διεθνή σκηνή, αλλά και να ε, μεριμνούμε έτσι ώστε αυτές τις εργασίες για τους ε, πολίτες μας όχι μόνο να διαφυλαχθούν, αλλά και να αναπτυχθούν, να πολλαπλασιαστούν. Αυτά είναι τα μελήματα τα οποία έχουν καθοδηγήσει και τις προτάσεις μας για τη μεταρρύθμιση, δηλαδή αποτελέσματα, στόχευση με αποτελέσματα, περιφερειακή και θεματική ανάπτυξη, με μεγάλη ευελιξία πρέπει να πω και πάντοτε αναφέρομαι στην ε, εικόνα ενός εστιατορίου το οποίο προτείνει ένα πολύ πλούσιο μενού αλλά από το οποίο μενού κανείς μπορεί να διαλέξει δύο ή τρία μόνο πιάτα και όχι 15. Αυτός είναι, αυτή είναι η προσέγγιση μας. με παράλληλα την αρχή της αίρεσιμότητας, της υπαγωγής σε προϋποθέσεις, έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά και σωστά αυτή η προσπάθεια. Σας ε, καλώ λοιπόν ε, να διατυπώσετε και εσείς από πλευρά σας να εκφράσετε την υποστήριξη σε αυτές τις προσπάθειες, ιδιαίτερα από τις χώρες που εισφέρουν, ε, που έχουν θετικό πρόσημο στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, πρέπει να πισθούν αυτές οι χώρες να μην προχωρήσουν σε περικοπές στις, στη συμβολή τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και πρέπει να βρούμε λύσεις, λύσεις για να λειτουργήσει να λειτουργεί η Ένωση με οικονομίες, ασφαλώς πολλές οικονομίες, αλλά εξυπηρετώντας πάντα το κοινό αυτό ευρωπαϊκό εγχείρημα το οποίο έχουμε ορίσει ως στόχο, στόχο μας με την Ευρώπη 2020 και γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια στον προπολογισμό. μείωση κλείνοντας ε, ότι αυτός ο πολιετής προπολογισμό σημαίνει αύξηση ε, εφόσον αποφασιστεί το 2012 θα καλύπτει τον, ε, την περίοδο μέχρι το 2020 και έτσι θα μπορούμε να προσφέρουμε και την σχετική ασφάλεια στον πολίτη για τα κονδύλια, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που μπορεί να περιμένει για την επόμενη ε, περίοδο αλλά όχι μόνο στον, πολίτη και οι διεθνείς αγορές θα πάρουν ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να ε, στηρίξει, να επενδύσει, να θέσει σε κίνηση την οικονομία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε οικονομική ανάπτυξη, εμπιστοσύνη και ευσιοδοξία για το μέλλον. Και ξέρετε όλοι οι οικονομολόγοι λένε ότι η οικονομία εξαρτάται κατά 50% τουλάχιστον από την ψυχολογική διάθεση. Άρα λοιπόν αν θέλουμε να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξία, πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερα ε, στου νέου επιχειρηματίε ότι μπορούν να έχουν ευκαιρίε, μπορούν να δημιουργήσουν. Έχουμε επί πράγματι μικροπιστώσει σε επίπεδο ευρωπαϊκό που μπορούν να αξιοποιηθούν από του νέου επιχειρηματίε. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει πρώτα να διατεθούν τα σχετικά κονδύλια. Γι' αυτό λοιπόν λέω τα μέσα υπάρχουν, οι λύσει υπάρχουν και πρέπει να προχωρήσουμε το, και η βούληση υπάρχει να προχωρήσουμε το δυνατό σε συνένεση, ε, σε κοινέ λύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα πρέπει και το, ευρω... το εθνικό επίπεδο κυρίε και κύριοι να κάνει ό,τι μπορεί. Uh, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον Επιβουλευτή, τον κύριο Κορνηλίου, να μας μιλήσει εκ μέρους ε, της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που ήρθα κάπως καθυστερημένα. Αλλά είναι και αυτό σημάδι ότι εργάζεται πάρα πολύ σκληρά η Προεδρία. Ήδη είχα και την πρώτη μου συνεδρίαση σήμερα και έπρεπε να τροποποιήσω την ώρα συνεδρίαση τη Κορεπέρη στι 10.30 γιατί θέλω να περιβρίσκομαι εδώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσκλησή σα, κύριε Επίτροπε, εξωτήμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την προσκλήση αυτή. Είναι τιμή μου και ευχαριστησή μου να βρίσκομαι εδώ και ήθελα να ευχαριστήσω και τους οργανωτές αυτής της σημαντικής εκδήλωσης ε, η οποία συμβάλλει στη στενότερη συνεργασία του Ευρωπαϊκού με Κοινοβούλια. Ο κύριος Στόχο της Κυπριακής Προεδρία είναι να εργαστεί προς μια καλύτερη Ευρώπη για μια ένωση η οποία θα σχετίζεται περισσότερο με τους πολίτες. Γι' αυτό υποστηρίζουμε θερμά κάθε προσπάθεια για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλίσουμε και να προωθήσουμε τον εκδημοκρατισμό στη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα αρμόδια όργανα, όλοι οι αρμόδιοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στι διαδικασίε λήψη αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα τη πολιτική που θα διαμορφώσει το μέλλον τη Ενωσή μα. Μένοντα στο τέταρτο μήνα τη Προεδρία μα, έχουμε πετύχει πολλά. Αλλά πρέπει να γίνουν και πολλά ακόμη. Η δική μας δέσμευση να εργαστούμε σκληρά είναι ιδιαίτερα ισχυρή και θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η κύρια προτεραιότητα τη Προεδρία μα είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει και να επιτευχθεί η πολιτική συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο πριν τα τέλη του 2012 η Προεδρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πετύχει μια ισορροπημένη και δίκαιη κατανομή στις κύριες τομείς πολιτικής βάσει της ποιότητας ε, των δαπανών και να διασφαλίσει ότι, τα προγράμματα, ότι έχουμε προγράμματα πραγματικής ευρωπαϊκής προσταμένης αξίας. Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία εργάζεται εντατικά για να πετύχει την μέγιστη δυνατή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για το νομοθετικό πλαίσιο των κοινών πολιτικών. Επιτρέψτε μου προς αυτή την κατεύθυνση να αναφερθώ περαιτέρω στο σημαντικό θέμα της πολιτικής συνοχής 2014-2020 οι συνεχιζόμενες συνέπειες ε, της ε, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης καθιστά απαιτητικό παρά ποτέ να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά του σπόρους. Η πολιτική συνοχή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επιτεύξη των κοινών μα στόχων, για τη μεγέθυνση και τι θέσει εργασία, ενώ διατηρεί το στόχο της για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή βάσει των θεμελιδών αρχών της ελληνική η διευκόλυνση μια εγκύρη συμφωνία ενό νομοθετικού πακέτου που θα διέπει ε, την πολιτική την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι μία από τι κυρίε προτεραιότητέ μα. Τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειε πρέπει να προετοιμαστούν ε, καλά πριν ξεκινήσει η νέα προγραμματική περίοδο, προκειμένου να υπάρξει ομαλή έναρξη τη εφαρμογή των νέων προγραμμάτων. Προ την κατεύθυνση αυτή, δεσμευόμαστε ω Προεδρία να βάλουμε τα δυνατά μας για την επιτεύξη της μέγιστης δυνατής προόδου στις διαπραγματεύσεις αυτές. Από τον Ιούλιο, η Προεδρία έχει ε, θέσει σε εφαρμογή ένα εντατικό πρόγραμμα στο Συμβούλιο για να ολοκληρωθούν όλα τα κρεμή θέματα της νομοθεσίας μέχρι τα τέλη του 2012. Φυσικά εξαιρούνται οικονομικά θέματα που ε, αφορούν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα θέματα που συζητούνται τώρα στο Συμβούλιο είναι μεταξύ άλλων η εδαφική ανάπτυξη, η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, χρηματοοικονομική διαχείριση και διαχείριση και συστήματα ελέγχου, καθώς και το πολύ σημαντικό κοινό στρατηγικό πλαίσιο που θα ε, διέπει την διατύπωση των νέων προγραμματικών εγγράφων. η σκληρή δουλειά ήδη απέφερε κάποιους καρπούς ε, την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, στο Συμβουλίο Γενικών Υποθέσεων. Μια προκαταρκτική συμφωνία αναμένεται να επιδευτεί στα κάποια από τα θέματα αυτά. Η πολιτική συνοχή επίση θα συμπεριληφθεί στην ατζέντα των Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του επόμενου μήνε, ε, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία στα υπόλοιπα ζητήματα. Ταυτόχρονα, Καλώς ορίζουμε και εκτιμούμε τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται μέχρι τώρα στο πλαίσιο της Περιφερειακής, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και Απασχόλησης που οδηγήσαν στην ψηφοφορία των ε, εκθέσεων που αφορούσαν ε, τις εκθέσεις σχετικά με το νομοθετικό πακέτο Περιφερειακής Πολιτικής. Η Προεδρία της Κύπρου δίνει συγκεκριμένη έμφαση σε μια στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο ως συνομοθέτη, αλλά και ως ένα κύριο εταίρο, προκειμένου να προωθήσουμε τον κοινό μας στόχο, κυρίως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Όπως γνωρίζετε πολύ εξημών, ε, ε, ε, έχει ξεκινήσει το τριμερής διάλογος για το νομοθετικό πακέτο. Η Προεδρία, μέρους του Συμβουλίου, διαπραγματεύεται θέματα που συμφωνήθηκαν ήδη υπό την Προεδρία της Δανίας βάσει της Γενικής Μερικής Προσέγγισης. Πιο συγκεκριμένα, για την τριμερής διάλογοι ξεκίνησαν ε, για τον ε, κανονισμό κοινών διατάξεων και για τον κανονισμό του Ευρωκοινωνικού Ταμείου το Νοέμβριο. Ε, θα ξεκινήσουμε τύπους τριμερείς διαλόγους για τον κανονισμό Ευρωπαϊκής Ταυτικής Συνεργασίας και για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης θέματα προγραμματισμού εξετάζονται ως πρώτη προτεραιότητα και από τα τρία όργανα. Η Προεδρία θέλει να πετύχει μια κανή συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων ε, θεσμών ε, στο θέμα του προγραμματισμού και έτσι θέλει να δοθεί μια ε, βεβαιότητα στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες για να προετοιμαστούν για τη νέα περίοδο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν για την επικοδομητική συνεργασία που διάπουν τις διαπραγματεύσεις σας μέχρι τώρα. Κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε, σε σχέση με τη σημερινή συζήτηση προς ένα κοινό στρατηγικό σχέδιο και σε συμβάσει εταιρική σχέση. Πριν να προχωρήσω, να εκφράσω την άποψη του Συμβουλίου, να μιλήσω για συμφωνίε εταιρική σχέση και όχι για συμβάσει εταιρική σχέση. Ε, και αυτό σημαίνει ότι δεσμεύεται ισχυρά το Συμβούλιο για να εφαρμοστούν τα νέα προγράμματα με πλήρη σεβασμό τη κυρία αρχή ε, τη εταιρική σχέση. Φυσικά, ε, υπό την επιφύλαξη των διαπραγματεύσεων με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτά τα νέα στοιχεία της πολιτικής συνοχής 2014-2020 είναι πάρα πολύ σημαντικά, καθώς θα παρατελέσουν τη βάση για την εφαρμογή μιας νέας γενιάς προγραμμάτων. Το Συμβούλιο καλωσορίζει την νέα προσέγγιση προτείνει Κομισιόν στο να ε, συμμετέχουν όχι μόνο τα διαθροτικά ταμεία αλλά και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ε, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Έτσι ε, θα έχουμε καλύτερο συντονισμό και συνέργειες μεταξύ των ταμείων αυτών αλλά και καλύτερε συνέργειε με άλλα μέσα πολιτική και μέσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο σήμερα εξετάζει την τροποποιημένη πρόταση τη Κομισιόν για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο να παράξει στην νομοθεσία τα πλέον σημαντικά στοιχεία που θα επιτρέψουν αποτελεσματικό συντονισμό και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό για την επιτεύξη των στόχων μα. Προ την κατεύθυνση αυτή, η Προεδρία της Κύπρου οργανώνει μια τύπο συνάντηση στις αρχές Νοεμβρίου στην Κύπρο όπου οι υπουργοί για την πολιτική συνοχή θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις ε, για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Όπως ήδη ανέφερα, σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς όπου τα αποτελέσματα της ε, οικονομικής κρίσης τα βλέπουμε καθημερινά άλλο ένα και πιο έντονα, πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των διαθεσιμών πόρων προκειμένου να πετύχουμε την ανάπτυξη και θέσει απασχόληση, δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να σκεφτούμε επί τη αποτελεσματικότητα και τη διακυβέρνηση τη νέα πολιτική συνοχή. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψει για το πώ τα νέα αυτά στοιχεία θα εφαρμοστούν επί τόπου διασφαλίζοντας ε, τα υψηλότερα πρότυπα ω προ την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα και ταυτόχρονα αντιμετωπίζοντα τι κυρίε προκλήσει ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καθώ και κάθε κράτου μέλου στην περιφέρεια. Πράγματι, το καθήκον μα είναι να παράξουμε το κατάλληλο πλαίσιο για τι περιφερειε για να μπορέσουν να βγουν από την κρίση. Κυρία Πρόεδρε, πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα και πάλι να εκφράσω την εκτίμησή μου που παρευρίσκομαι εδώ σήμερα. Επαναλαμβάνω την έκκληση της Προεδρίας για συνεργασία και εταιρική σχέση στις προσπαθίες μας για μια καλύτερη Ευρώπη. Φυσικά αυτή η έκκληση αναφέρεται και στα εθνικά κοινοβούλια που στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής έχουν το προνόμιο να έρχονται σε στενή επαφή με ε, τις τοπικές αρχές και να ενδυναμώνουν, να συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της ε, πολυδιακυβέρνησης, μιας ε, πρακτικής που έχει επιφέρει πραγματικά προσθεμένη αξία για την πολιτική συνοχή στα τελευταία χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Να πω και εγώ κάτι τελευταίο Είμαι από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόεδρος ε, των ε, διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου και πρέπει να σας πω ότι παρότι έχουμε σημειώσει πρόοδο, πολλά ακόμη από να γίνουν. Συμφωνώ μαζί σας κύριε Πρέσβη και εμείς θα θέλαμε οι διαπραγματεύσεις να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Και ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεισφέρει να το πετύχουμε το στόχο αυτό. Τώρα, μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Να πω όμως πρώτα δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο Επίτροπος ε, έχει να συζητήσει με ε, τον Επίτροπο Αλμούνια, ένα θέμα που αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο ε, και για τα οικονομικά ζητήματα, γι' αυτό και δεν μπορεί να είναι μαζί μας πια. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια έχετε ένα φάκελο μπροστά σας και έχετε και αυτές τις κάρτες που σας δίνω, που ουσιαστικά είναι η κάρτα που πρέπει να συμπληρώνετε για να λάβετε το λόγο. Θα ήθελα να ξέρω ε, λίγο πολύ ποιοι θέλουν να μιλήσουν για να δω πώς θα οργανώσουμε και το χρόνο μας και το χρόνο αγόρευσης. Ο Νίκολας Μάρτιν, ο αναπληρωτής Γενικός ε, Διευθυντής της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΡΕΓΙΟ της Ευρωπαϊκής Πολιτικής αντικαθιστά τον Επίτροπο που όπως είπα έπρεπε να φύγει και είναι ο αρμόδιος για τις διαπραγματεύσεις από πλευράς κομισιών. Έχουμε δύο συναδέλφους μαζί μας προερχόμενους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, τον κύριο Ράινερ Ρόμπρα ο οποίος ε, είναι υπουργός ε, και επικεφαλής της ε, καγκελαρίας της Αξονίας Άνχαλτ. Είναι και μέλος της γερμανικής Bundesrat. Έπειτα έχουμε τον κύριο Λάιαμ Τουόμι, που είναι ότι πρόεδρος Τώρα πώς θα το προφέρω αυτό. Έχετε εδώ στα Ιρλανδικά 100 φωνήεντα και, και σύμφωνα και προφέρετε το ένα από αυτά. Δεν θα το λέω. Τέλος πάντων είστε υπεύθυνο για τα οικονομικά ζητήματα, είστε αντιπρόεδρος Επιτροπής Μεταρρυθμισής. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρόμπρα. Ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι, χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω ενώπιον του εκεκριμένου σας κοινού. Ίσως να μην αισθάνονται ικανοποιημένοι πολλοί από τους εδώ παρόντες με τα αποτελέσματα της στρατηγικής Λισαβόνας. Ε, μέχρι το 2010 έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία του κόσμου. Το στόχο αυτόν τον έχουμε χάσει. Έχουμε αποτύχει εκτρά και δεν θέλω να ρίχνω αλάτι στις πληγές, δεν θέλω να ξύνω πολλέ πληγές, αλλά θέλω να πω ότι μπορούμε όλα τα κράτη μαζί και μαζί με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίσουμε να ε, ορίσουμε νέα ορόσημα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και την υλοποίηση ευφύους, βιώσιμης και ανοιχτή σε όλους ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ο στόχος της στρατηγικής Λισαβόνας είχε ως βάση μια σωστή μεταρρύθμιση των δομών, ανάπτυξη, καινοτομία, έρευνα, κατάρτιση, δεξιότητες, διαβίου βάση, ε, μάθηση, εξυγίανση των δημοσιονομικών τομείς δηλαδή που πάντα χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα ακόμη για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, των δημογραφικών αλλαγών, για να διασφαλίσει θέσεις εργασίας, για να ενισχύσει το επίπεδο ευημερία. Αλλά η στρατηγική της Λισαβόνας δεν προσέφερε το κατάλληλο μηχανισμό, τα κατάλληλα μέσα δηλαδή για την προαγωγή των στόχων αυτών και την καταπολέμηση εξυπαρχής της κρίσης. Εξού και θεωρώ ότι είναι σωστό και συνεπές το να διατυπώνει κανείς το αίτημα για μια σαφέστερη διατύπωση των στόχων της στρατηγικής Λισαβόνας και την ε, εξασφάλιση, την αξιοποίηση καλύτερα όλων των μέσων που είναι απαραίτητα για την υλοποίησή της. Η Επιτροπή έχει δραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, λισαβονοποίηση όπως ονομάζεται, ε, η λισαβονοποίηση παραδείγμα των εθνωτικών ε, ταμείων έχει οδηγήσει σε πολύ σημαντικές ενισχύσεις των ποσών 228 δισεκατομμύρια από το 7 στο 13, ενίσχυση των ποσών για την ανάπτυξη, για τις επιχειρήσεις και έτσι η λύσεις που προτείνονται, οι ιδέες για μια ανεπτυξιακή στρατηγική για την περίοδο έως το 2020 δεν ε, προσπαθούν να διερευνήσουν παρθένο έδαφος είναι ήδη γνωστές λύσεις. Εμείς, ε, τη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, η Σαξονία Άνχαλτ, έχει υποφεληθεί από, τις, ε, από την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από, την, ε, από τους στόχους της συνοχής βρισκόμαστε πλέον για την επόμενη περίοδο στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 μπορεί να καταστεί αποτελεσματική και επιτυχής μόνο εάν ο στόχος της συνοχής προσδιορίσει τους κεντρικούς Στοχό στόχους, της κεντρικές προτεραιότητες με τις ανάγκες, σε συγκερασμό με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Η εταιρική σχέση στην διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική αρχή, η πολιτική συνοχή πρέπει να αναπτυχθεί και να, να γίνει αποδεκτή από τον πολίτη της Ευρώπης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμοποίηση και η συμπλήρωση των σχεδίων, όχι αντικατάστασή τους αλλά συμπλήρωσή τους με, την, με τις προτάσεις των πολιτών η στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι η πραγματικά ουσιαστική εκδοχή του τι σημαίνει Ευρώπη για το 2020. Είναι ένα όραμα το οποίο όμως θα αποτύχει αν δεν έχουμε την μόρφωση, την κατάρτιση, την βιωσιμότητα, το επίπεδο της απασχόλησης που θα μπορέσουμε να ελοπίσουμε στην κάθε περιοχή επιτόπου δηλαδή και ως εκ τούτου η, πολιτική συνοχή δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί επουδενή και αυτό το λέω και με παράδειγμα τη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα. Έχουμε μεγάλες προκλήσεις προκλήσεις που έχουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε βράχη και μέσο πρόθεσμα. Έχουμε καθυστέρηση σε ανάπτυξη, δυσκολίες στη δημογραφική ανάπτυξη, εντά, ε, χάσμα μεταξύ προσδοκιών ανάπτυξη μηχανικής και ε, γεωργικής, ε, απουσία εργατικού δυναμικού σε ένα μεγάλο βαθμό, προβλήματα ως προς την ε, ε, που προσφέρουμε στα παιδιά μας και βέβαια το πρόβλημα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, το, το οποίο βρίσκεται υπό την ομπρέλα της συνταγματικής απαγόρευσης που έχουμε στη Γερμανία για απόκτηση χρέους από ένα κρατήδιο. Κανένα κρατήδιο στη Γερμανία δεν μπορεί να χρεωθεί, να χρεώσει τον προπολογισμό του με χρέους. Ε, όμως έχουμε από την άλλη μεγάλες ευκαιρίες να δράξουμε, έχουμε πολλά θετικά στοιχεία να διαφυλάξουμε και μπορούμε νομίζω να λάβουμε αποφάσεις στοχευμένα, να τις γρήγορα και να διορθώσουμε το ταχύτατο δυνατό τις ε, καθυστερήσεις, τα προβλήματα στην υλοποίηση που έχουν εντοπιστεί. Αυτό για τους πολίτες της ε, ιδιαίτερης μου πατρίδας του κρατηδίου μου είναι σημαντικό, όπως είναι σημαντικό για κάθε πόλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα θέλω να επισέλθω στα επιμέρους προβλήματα, όπως όλα τα κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, τα ανατολικά κρατήδια της Γερμανίας, παρουσιάζει η Σαξονία Άνχαλτ ε, καθυστέρηση, προβλήματα ως προς την ε, εξισορρόπηση των ε, δαπανών και των εσόδων και μεγάλες διαφορές ισοδηματικές στον πληθυσμό που προχωρεί και από τις τελευταίες εκθέσεις ε, που εντοπίζουν ε, πρόβλημα ε, στην οικονομική δύναμη, στην αγοραστική δύναμη δηλαδή των πολιτών. Βλέπουμε δυστυχώς ότι έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά 2 με 3% αυτή η διαφορά αγοραστικής δύναμης μεταξύ των ανατολικών και των δυτικών κρατοδίων της Γερμανίας. Δεν υπάρχουν επίσης επενδύσεις ε, σημαντικές από μεγάλες επιχειρήσεις στις περιοχές μας. Δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, τα νέα λεγόμενα γερμανικά κρατήδια έχουν μεγάλες ε, προκλήσεις να αντιμετωπίσουν με τη γύρανση του πληθυσμού και την έλλειψη εργατικού δυναμικού από πλευράς δηλαδή δημογραφικών ε, προκλήσεων δεν υπάρχει περιοχή της Ευρώπης που να έχει πληγεί τόσο πολύ και από την μετανάστευση, την έξοδο δηλαδή των πολιτών, αλλά και τη γύρανση του πληθυσμού όσο τα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας. Αυτό σημαίνει βέβαια και χαμηλότερη ε, είσοδα, έσοδα φορολογικά και κοινοτικά στους Δήμους και τις κοινότητες. Έτσι, ε, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα χρειάζεται και καλύτερη διαχείριση των ανθρωπινών πόρων και βελτίωση των οικονομικών των εισόδων. Άρα λοιπόν όλα τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό ε, στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να αξιοποιηθούν Δυνάμε το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σαξονία Άνχαλτ, την Ανατολική Γερμανία και όλες αυτές τις περιοχές οι οποίες πλέον δεν υπάγονται στους στόχους της συνοχής χρειάζεται μια μεσοπρόθεσμη πιστεύω διάθεση κονδυλίων με ένα σύστημα ασφαλείας όπως έχει πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο στα δύο τρίτα των, ε, της που έχουν αυτή τη στιγμή και ένα περιθώριο ακόμη για την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προβλημάτων. Αυτό το λεγόμενο δίκτυο ασφαλείας μπορεί να έχει τεράστια σημασία και να φέρει πολύ σημαντικές εξελίξεις στην, ε, στα κρατήρια της Γερμανίας. Αυτές οι προτάσεις και τα αιτήματα δεν είναι σε αντίθεση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 των αντίων. θα την υλοποιήσουν πολύ ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά. Και έτσι ένα ποσοστό κεντρικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του 40% όπως έχει προσδιορισμηθεί, Δεν ξέρουμε αν είναι μια καλή λύση. Εμείς έχουμε ήδη με το 30% που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή ως ποσοστό πρόβλημα απορρόφησης πόρων και άρα ένα τέτοιο ποσοστό, τόσο υψηλό ποσοστό δεν ξέρω αν θα ήταν αποτελεσματικό. Θα οδηγούσε τελικά σε ακόμη μεγαλύτερη περικοπή των πόρων που είναι διαθέσιμοι για επενδύσεις στις επιχειρήσεις μας. Επίσης, χρειάζεται να προσδιοριστούν και έξω από τη μέχρι τώρα στενή θεματολογία νέοι στόχοι για επενδύσεις, για μεγάλες επενδύσεις. Ή μερικές και γενικές. Ε, κατευθύνσεις που υιοθέτησε το Συμβούλιο τον Ιούνιο δίνει, δίνουν νομίζω πολύ σημαντικές προοπτικές βελτίωσης για τις περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλουν στον τριμερή διάλογο στην ε, ε, έτσι περαιτέρω βελτίωση των προτάσεων των κρατών μελών. Και για να κλείσω, έχουμε μια τριπλή πρόκληση. Έχουμε τα, προγρά... έγγραφα προγραμματισμού, έχουμε τις ε, εταιρικέ συμβατικές σχέσεις και τις ε, τοπικές αρχές, όπως έχουμε στη Γερμανία το σύστημα των ε, τοπικών κοινοβουλίων, ένα, μια τριαδική δηλαδή προσέγγιση με βάση την οποία θα αναπτύξουμε αυτές τις προσπάθειες στη Γερμανία. Οι εταιρικέ συμβατικές σχέσεις μερικές φορές χαρακτηρίζονται ως κακή λύση. Εγώ θα ήθελα όμως σε αυτό και από την εμπειρία που έχουμε στο κρατήδιο της ε, Σαξονίας Άνχαλτ να υπογραμμίσω ότι δεν είναι σωστό αυτό, γιατί πρέπει να έχουμε την ε, συνεργασία, την εταιρική σχέση με τους ενδιαφερόμενους, με τους άμεσα εμπλεκόμενους, ε, ακόμη και για την υλοποίηση του στόχου της αποδεξιμότητας της νομιμοποίησης δηλαδή των σχεδίων που προβάλλουμε. Η δε ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών δεν θα πρέπει να υποτιμάται. Πρόκειται για μια ε, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που λαμβάνει η χώρα διαρκώς μέσα από αυτές τις συμβατικές εταιρικέ σχέσεις, αλλά βέβαια ο κίνδυνος θα ήταν ε, μέσα από το διαρθρωτικό ταμείο να τυποποιηθούν τόσο πολύ οι σχέσεις, ε, το πλέγμα των σχέσεων να μετατραπεί σε τόσο γραφειοκρατικό, ώστε να μην έχει πια τη δυναμική και την παραγωγή αποτελέσματος. για την περίοδο 2014-2020 θέλουμε μία παρακολούθηση των προγραμμάτων που έχουν προβλεφθεί με ε, workshops, με εργαστήρια, καταρχάς για την ε, καινοτομία και την συνεργασία στην διεθνή ανάπτυξη, δεύτερον για τις ε, δημογραφικές αλλαγές, την αποχώρηση, ιστορική μετανάστευση δηλαδή, τρίτον για την κατάρτιση, εκπαίδευση μάλλον και μέρημνα για τα παιδιά, Τέταρτον, ε, μετανάστευση, ε, αποδοχή των, ε, του αλλοδαπού και προγράμματα τέτοια, τα οποία ήδη έχουμε αναπτύξει στην προηγούμενη περίοδο και που αποτελούν ιδιαίτερα σε ένα κράτος ε, ομοσπονδιακό προϋπόθεση ή εξασφαλίζουν καλύτερα την προϋπόθεση της νομοποίησης, δημογραφικής ε, νομοποίησης με τη συμμετοχή των διαφορών οικονομικών παραγόντων, όπως προγράμμισε και ο Επίτροπος ε, Ντεχάν, τα προγράμματα αυτά, ε, ο Επίτροπος Χάν, τα προγράμματα αυτά θα ισχύσουν έως το 2020 και θα διαμορφώσουν την περίοδο αυτή. Τα θέματα τώρα της κοινοβουλευτικής συμμετοχή στη διαμόρφωση των προγραμμάτων αυτών, συμμετοχή των κοινοβουλίων. Δεν έχουν επιληθεί. Εμεί από τη Σεξονία Άνχαλτ προσπαθούμε διαρκώ ε, να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή των βουλευτών στον διάλογο αυτό και ενημέρωση του τοπικού κοινοβουλίου για την εξέλιξη των ε, προγραμμάτων. Και με την ε, εντονότερη διασύνδεση που προβλέπεται τώρα στη νέα, στη νέα γενιά προγραμμάτων, στον κύκλο της Ευρώπης 2020, ε, στρατηγική αυτή δηλαδή, βλέπουμε νέες δυσκολίες, ότι δηλαδή τα προγράμματα μεταρρύθμισης, τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης με ειδικέ προτάσεις για τα κρατήδια και με σημαντικές ε, προϋποθέσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Όταν προχωρήσω αυτά τα προγράμματα, πώς θα είμαστε βέβαιοι ότι αρκεί η αρκεί αυτός ο προγραμματισμός και είναι παρκός και δημοκρατικά νομοποιημένος. Χρειάζεται οπωσδήποτε να προβλεφθεί μια περίοδος κατά την οποία με συμμετοχή των, των τοπικών κοινοβουλίων θα συζητηθούν και θα ενσωματωθούν στην εσωτερική τάξη του κρατηδίου για να γίνουν αποδεκτά τα προγράμματα αυτά και οι συμφωνίες αυτές. που οπωσδήποτε έτσι θα έχουν καλύτερη αποδοχή. Αυτή τη στιγμή δεν έχω λύσεις καταληκτικές να προσφέρω, αλλά καλό τους πάντες να ε, διατηρήσουν σε υψηλή προτεραιότητα το ζήτημα της συμμετοχής των κοινοβουλίων. Κυρίε και κύριοι, μιλάμε πολλές φορές εδώ στην Ευρώπη αυτήν την εποχή για κρίση, ακόμη και για αποτυχία της πολιτικής έχουμε ένα από τα μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες να αντιμετωπίσουμε αυτή την εποχή και θα ήθελα να πω ότι και εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφυλάξει την δύναμη της, την ισχύ της να προχωρήσει και να αλλάξει. Η πολιτική συνοχή είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαμόρφωση της απασχόλησης, ε, της ε, ανάπτυξης Τη ευημερία και θέλουμε οπωσδήποτε εμεί και από τη Σαξονία Ανχάλτ να διαφυλάξουμε αυτή την δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα είναι πιστεύω και η ισχυρότερη συμβολή στην υλοποίηση του στόχου της Ευρώπης 2020. Σα ευχαριστώ θερμά. Thank you. Uh, thank you indeed. Σας ευχαριστώ θερμότατα που μοιραστήκατε μαζί μας ε, και ε, κάποια ιδιαίτερα στοιχεία για την ε, Σαξονία Άνχαλτ που θα μας βοηθήσουν και μας και να παρακαλέσω τώρα τον κύριο Λίαμ Τάμι να μας παρουσιάσει τα Ιρλανδικά θέματα. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Περιφερειακή Πολιτική που διοργάνωσε τη σημερινή διακοινοβουλευτική συνάντηση που νομίζουμε ότι ασχολείται με ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα. Πρέπει να ε, πούμε ότι η πολιτική συνοχή είναι μια επιτυχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στο επίκεντρο τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αλληλεγγύη. Και παίζει μείζωνα ρόλο για τη των οικονομικών, κοινωνικών ανισοτήτων και την αύξηση της συνοχής σε μια Ευρώπη 500 εκατομμυρίων κατοίκων και 27 κρατών μελών και 271 ε, περιφερειών. Δεν θα πρέπει λοιπόν τη συνοχή να την υποτιμούμε. Μιλώ ε, από προσωπική εμπειρία και πρέπει να σας πω ότι η χρηματοδότηση συνοχής έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για την ανάπτυξη της Ιρλανδικής οικονομίας. Οι μεταφορές πιστώσεων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ήταν κάτι πολύ σημαντικό που έδωσε τη δυνατότητα ε, στην Ιρλανδία και στις περιφέρειές της να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Όπου και αν κοιτάξει κανείς στη χώρα μου μπορεί να δει ε, ότι ε, στις διάφορες πινακίδες των έργων ε, βλέπουμε χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Έχουμε ωφεληθεί λοιπόν από κονδύλια των διευθυντικών ταμείων. Πρέπει να σας πω ότι η ε, είναι μία από τις επιτυχημένες ιστορίες που έχει να κάνει τα διευθυντικά ταμεία. Βλέπουμε όμως ότι και άλλες χώρες μπορούν να αποφεληθούν από αυτά και μάλιστα έχουν σταλεί εκπρόσωποι των κρατών αυτών ε, μελών στην Ιρλανδία για να δουν ε, και να αντλήσουν θετικές εμπειρίες. Τώρα, έχουμε μια οικονομική ύφεση αυτή την περίοδο. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις για την ολοκληρωμένη πολιτική συνοχή. Θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχή θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να πετύχουμε τις προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και πρέπει να προωθήσουμε την ευφυή βιώσιμη ανάπτυξη για όλους που δημιουργεί την βασική κατεύθυνση για τη μελλοντική πολιτική. Πιστεύουμε ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εστιάζονται στην απασχόληση, την έρευνα και καινοτομία, την παιδεία, την καταπολέμηση της φτώχειας, την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια. Θα γνωρίζετε ότι πέρυσι δημοσίευσε η Κομισιόν τις προτάσεις της για τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης για την περίοδο 2014-2020. Προτάσεις της Κομισιόν είναι 376 δισεκατομμύρια ευρώ να δοθούν σε μέσα και εργαλεία πολιτικής συνοχής και να αυξηθούν ε, τα κονδύλια τα οποία προβλέπονταν για την προηγούμενη περίοδο 2007-2013. Βέβαια όλα αυτά ε, μπορεί να μειωθούν λόγω των πιέσεων που θα ασκηθούν για μείωση του συνολικού προπολογισμού στι διαπραγματεύσει τη τριμερή. Τον Οκτώβριο παρουσίασε και κάποια άλλα στοιχεία η Κομισιόν ε, και εμείς ε, θα συμμετάσχουμε και στις διαπραγματεύσεις και στις συνομιλίες για τη διαμόρφωση του μελλοντικού πακέτου συνοχής. Ο Υπουργός Δημόσιων ε, Δαπανών και Μεταρρύθμισης που είναι υπεύθυνο για τις πολιτικές συνοχής ήδη έχει συζητήσει με τους ομολόγους του σε μια άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Συνοχής τα σχετικά επί Πολωνικής Προεδρίας και σε Υπουργείο των, και σε συνεδρίαση μάλλον του του Δεκεμβρίου του προηγούμενου, ενώ συμμετείχε και στην κοινοβουλευτική συνέλευση που συνάντησε στι 3 Οκτωβρίου την Κομισιόν και συζήτησε τα σχέδια της Ιρλανδική Προεδρίας. Και είχαμε και μια διμερή συνάντηση με τον Επίτροπο Χάν τον επόμενο μήνα μάλιστα το Επίτροπο θα επισκεφτεί την Ιρλανδία. Ο Υπουργό συνάντησε εκπροσώπους του Κοινοβουλίου όταν πρόσφατα επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες και προσβλέπει να συναντήσει και εκπροσώπους της αντιπροσωπείας ε, της ε, Επιτροπής σας που θα έρθουν ε, στις 28 έως 20 Νοεμβρίου 2012 στο Δουβλίνο και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συζητούμε την γενική προσέγγιση. Έχουμε καταλήξει σε κάποια ε, στοιχεία του διαπραγματευτικού κουτιού, αλλά ε, αναμένονται περαιτέρω συζητήσει για τι διαρθρωτικέ δράσεις στην αρμόδια ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Το 2012 έγιναν εντατικέ διαπραγματεύσει σε Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο για το πακέτο συνοχή. Η θέση τη Ιρλανδία στι διαπραγματεύσει αντικατοπτρίζει το μεγάλο αντίκτυπο που έχει και είχε η χρηματοδότηση συνοχή σε πολύ σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά προγράμματα σε ολόκληρη την Ιρλανδία. Η χρηματοδότηση για το 2014-2020 πρέπει να παραμείνει στα ίδια επίπεδα για να μπορέσει να ανακάμψει η Ιρλανδία δεν μπορούμε να έχουμε ένα μέγεθος για όλους και γι' αυτό θεωρούμε ότι καλύτερο θα ήταν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να έχουν την απαιτούμενη ευελιξία για να επιλέγουν τις προτεραιότητές τους ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν ε, στις χώρες περιφέρειες και τα ε, σχετικά των εθνικών μεταρρυθμιστικών τους σχεδίων. Με αυτή την προσέγγιση οι περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν ε, τα μέσα, τις πολιτικές που θα μπορούν να τα αποκριθούν στις ιδιαίτερε τους ανάγκες και θα παράσχουν επίσης, θα προβλέψουν μάλλον την ισχυρότερη συμμετοχή και ε, ανάληψη όλων αυτών των πρωτοβουλειών και επιτόπου. Πρέπει να προστατεύσουμε την διαφοροποίηση στην Ευρώπη. Οι περιφέρειες έχουν πάρα πολύ μεγάλες ε, ε, διαφορές, έχουν όμως και ευκαιρίες, έχουν και ανάγκες διαφορετικές. Η πρόταση της Κομισιόν για ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο και για τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης έχουν τη δυνατότητα να ε, οδηγήσουν σε μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα, συντονισμό, συνεκτικότητα και συνέργεια μεταξύ των διαφόρων ταμείων συνοχή, αλλά και για την ανάπτυξη της υπαίθρου και για την αλληλευτική πολιτική. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητα θα ληφθούν επαρκώ υπόψη και ότι τα διοικητικά βάρη δεν θα αυξηθούν περαιτέρω. Τέλος, Εν, εν συντομία θα ήθελα να σχολιάσω την επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία που έχει ως στόχο να διευκολύνει την επίτευξη πρόοδου για την πολιτική συνοχής. Ίσως ε, οι διαπραγματεύσεις ε, στο επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών για την ολοκλήρωση του πακέτου συνοχής να πέσουν στο εξάμεινο της δικής μας Προεδρίας. Και επίσης και η συζήτηση επί του όλου νομοθετικού πακέτου και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση για την κυβέρνησή μας. Προσβλέπουμε όμως και είμαστε πεπισμένοι ότι θα πετύχουμε, θα αφοσιωθούμε πλήρως, θα εφαρμόσουμε πλήρως και τη διαδικασία συναπόφασης και θα συνεργαστούμε πλήρως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να συγχαρώ τη Δανική και την Κυπριακή Προεδρία για το έργο που επιτέλεσαν και την πρόοδο που σημείωσαν σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που ε, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το πακέτο συνοχής. Εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω και θα συμμετάσχω ενεργά και στην συζήτηση που θα επακολουθήσει. Με βέβαιος ότι ο γύρος ερωταπαντήσεων που θα ακολουθήσει θα είναι πάρα πολύ επικοδομητικός για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ε, διαβεβαιώσω ότι ε, όλα τα έχει αναλάβει η Κυπριακή Προεδρία και θέλω να σας πω ε, ότι θα, είχαν ολοκληρωθεί όλα από την, μέχρι την Ελλαδική Προεδρία, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Αν ε, δεν μου ζητήσουν κι άλλοι το λόγο αυτή τη στιγμή, μπορώ να σας δώσω πέντε λεπτά. Και θέλω να ζητήσω από όλου να σεβαστείτε το όριο αυτό το χρονικό των πέντε λεπτών και να σας ενημερώσω ότι θα έχουμε δύο εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με αυτή τη σειρά λοιπόν θέλουμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Καταρχήν ε, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο κυρίος Δημήτρης Αμπαζιώτης. Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην τόσο σημαντική συνάντηση με θέμα την πολιτική συνοχή από το 2014 το 2020. Επίσης να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης ε, η οποία σίγουρα ε, βελτιώνει πολύ την συνοχή ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Κυρίες και κύριοι, κάθε 7 χρόνια τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύονται επί διετία τον επταετή του προϋπολογισμό, γνωστό και ως πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρόκειται κατά γενική εκτίμηση για μια από τις δυσκολότερες και πλέον πολύπλοκες διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ευνόητες πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είναι γνωστό πω η πολιτική τη οικονομική και κοινωνική συνοχή κατοχυρώνεται στι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί βασική αρχή τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και το στόχο και προπόθεση τη ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά στην ΟΝΕ. Τα τελευταία 20 χρόνια η υλοποίηση των πολιτικών της συνοχής δεν ωφελεί μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, αλλά και τα κράτη-μέλη που είναι καθαρή συνεισφορή του κοινοτικού προπολογισμού, είτε μέσω στήριξη περιφερειών του με προβλήματα υστέρηση, είτε έμεσα με τη δραστηριοποίηση των εταιριών του και την αύξηση των εξαγωγών του στι χώρε τη συνοχή. Υποστηρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια φιλόδοξη πολιτική συνοχή, δεδομένου ότι προσφέρει ολοκληρωμένη προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη. Διαφωνούμε με τοποθετήσει που αναδεικνύουν διακρίσει μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών η πολιτική συνοχή αφορά όλε τι περιφέρειες του συνόλου των κρατών μελών, επιτρέποντα σε αυτέ να υποστηρίξουν τόσο το στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξή του, όσο και την κοινωνική συνοχή των περιφερειών του. Η Ελλάδα, με δεδομένη την μεγάλη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει, καλείται να λειτουργήσει σε ένα δυσμενέ για αυτή πλαίσιο, λόγω τη ένταξη των φτωχότερων χωρών και του γενικότερου περιοριστικού δημοσιονομικού κλίματο. Από το σύνολο των πολιτικών του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου άμεσης προτεραιότητας για την ελληνική πλευρά είναι η πολιτική συνοχή, η κοινωνική αγροτική πολιτική και η πολιτική μετανάστευση. Οι προτάσει μα για τα σημαντικότερα επιμέρου ζητήματα του διαπραγματευτικού πακέτου για την πολιτική συνοχή είναι οι εξή. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τα προτινόμενα στατιστικά στοιχεία για τη μεθοδολογία κατανομή των κονδυλίων τη πολιτική συνοχή, επειδή είναι τη περίοδου 7 έω 9, θεωρούμε πως αποκλίνουν σημαντικά από την τρέχουσα πραγματικότητα καθώς δεν αποτυπώνουν την αρνητική επίπτωση της ύφεσης και της βαθιάς οικονομικής κρίσης. Συνεπώς σε μια κρίσιμη καμπή για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατανομή των κονδυλίων της συνοχής βασίζεται σε μια ξεπερασμένη εικόνα της οικονομίας των κρατών μελών και των περιφερειών τους υποστηρίζουμε ότι το μέγεθο τη πτώση του ΑΕΠ σε σχέση με την ταυτόχρονη άνοδο των ποσοστών ανεργία εντό των κρατών μελών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν θα γίνουν τελικέ ρυθμίσει στι μεθόδου κατανομή πόρων τη συνοχή. Δεύτερον, υποστηρίζουμε ότι η μακροοικονομική αιρεσιμότητα δεν πρέπει να συνδέεται με τον κοινοτικό προπολογισμό, ο οποίο αποτελεί κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τυχόν επέκταση. There is a request from interpreters that you slow down a little bit. Okay τυχόν επέκταση της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας πέραν του Ταμείου Συνοχής σε όλα τα διαφορετικά ταμεία αποτελεί διπλή επιβράδυνση για τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη-μέλη, δεδομένου ότι ήδη προβλέπονται ποινές για τα κράτη-μέλη τόσο στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, όσο και στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η επιβολή περαιτέρω ποινών που πλήττουν άμεσα τις περιφέρειες για δυναμίες σε εθνικό και όχι σε περιφερειακό επίπεδο λειτουργεί στην πράξη αντιαναπτυξιακά οδηγώντας σε ένα φαύλο κύκλο ύφεση. Τρίτον, η Ελλάδα υποστηρίζει την αύξηση ή τουλάχιστον τη διατήρηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης της τρέχουσας περίοδου και στη νέα δημοσιονομική περίοδο. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει να είναι ανάλογα με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του κράτους μέλους και να μην καθορίζονται με οριζόντιο τρόπο σε περιφερειακό επίπεδο σε σχέση με τα εισοδήματα των περιφερειών τους. Επίσης, υποστηρίζουμε την πρόβλεψη αυξημένης συγχρηματοδότησης κατά 10% για κράτη-μέλη που λειτουργούν εντός του μηχανισμού στήριξης μέσω διαδικασιών γρήγορης ροής των κοινοτικών κονδυλίων η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί σημαντική βοήθεια προς την κατεύθυνση ανάκαμψης των κρατών μελών που πλήττονται περισσότερο από τη δυσχερή οικονομική κρίση ενώ παράλληλα έχει προστιθέμενη αξία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτον, διαφωνούμε με την διασύνδεση του ύψους των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής καθώς και της προχρηματοδότησης των έργων στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής με το θέμα των εναπομενουσών πιστώσεων προς αποπληρωμή το θέμα των πιστώσεων αυτών προς αποπληρωμή οφείλεται σε ανεπαρκείς ετήσιες πιστώσεις πληρωμών και αποτελεί αντικείμενο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και όχι του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Πέμπτον, υποστηρίζουμε την επέκταση του δικτύου ασφαλείας που προβλέπει την διατήρηση των δύο τρίτων των πόρων των περιφερειών εξερχομένων στόχου 1 και τις περιφέρειες στατιστικής σύγκλησης. Στο ζήτημα αυτό είναι κρίσιμη σημασία για την Ελλάδα, δεδομένου ότι περιφέρειε στατιστική σύγκληση όπω η περιφέρεια Αττικής, λόγω αυξημένου ΑΕΠ, θα κατατάσσεται πλέον μεταξύ των πιο εύπορων περιφερειών. Έτσι η περιφέρεια Αττικής αναμένεται να λάβει σημαντικά μειωμένου πόρους σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο. Τέλος, θεωρώνταμε ότι επιλέξιμε στην ενδιάμεση κατηγορία θα πρέπει να είναι και οι περιφέρειες με γεωγραφικέ ιδιαίτερότητε δηλαδή γεωγραφικά μειονεκτήματα όπως τα νησιά. Ειδικότερα στην κατεύθυνση αυτή υποστηρίζουμε τη μόνιμη ένταξη όλων των νησιωτικών περιφερειών οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο στόχο σύγκλησης, στον ενδιάμεσο στόχο της πολιτικής συνοχής, ανεξαρτήτως επίπεδου του ΑΕΠ. Η συμπερίληψη του νησιώτικου χώρου στα διευρωπαϊκά δίκτυα και στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, συνδέοντας την Ευρώπη και την αναγνώριση του κόστους της νησιωτικότητας. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης, στην Ευρώπη με δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις, η πολιτική συνοχής οφείλει και πρέπει να θέτει πιο φιλόδοξους στόχους. Διαφορετικά, κράτη-μέλη και περιφέρειες σε ύφεση δεν θα είναι δυνατόν να προχωρήσουν σε αναπτυξιακές επενδύσεις λόγω ουσιαστικά α, απόλυτης έλλειψης εθνικών πόρων και συνεπώς δεν θα μπορούν να εξέλθουν από αυτήν. Υπό τις παρούσες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και την περίοδο ύφεση που διανύουμε, η επίδειξη αλληλεγγύης και οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη της οικονομίας, την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας είναι περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ. Ιδιαίτερα για κράτη που βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα της οικονομικής κρίσης όπως η χώρα μου η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στη Σουηδία. Την κυρία Κρίστεν Ερίευτε. Τον κύριο. Με συγχωρείτε, νόμιζα ότι ήταν Χριστίνα το κρίστε στα Σουηδικά. Θα το δεχτώ, θα το δεχτώ, λέει ο μιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Σουηδικά, καθώς ε, έχω την ευκαιρία αυτή σήμερα. Η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή ανήκει στους ε, κυρίους στόχους της κυβέρνησης ε, στο δημοσιονομικό πλαίσιο αυτό. Σημαίνει ότι δεν θέλουμε να τροποποιηθούν ε, οι ευρωπαϊκές πληρωμές. Τώρα έχουμε αυτές τις διάφορες κατηγορίες ΑΕΠ από το 95-97% του μεσόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε ότι θα πρέπει, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο χρονικό αλλά και στο πεδίο εφαρμογή. Ε, η Επιτροπή υποστηρίζει το στόχο μείωση ε, του κατοφλίου σε σχέση με το ΑΕΠ. Σε πολλέ περιπτώσει αυτό σημαίνει προσαρμογή στην ε, πραγματική ικανότητα και έχει και ένα αποτέλεσμα περιορισμού του προπολογισμού. Τώρα, η ακριβή διατύπωση και πώ αυτό μπορεί να θίξει τα μεμονωμένα κράτη-μέλη, ίσω είναι κάτι που θα πρέπει να αναλυθεί. Η Επιτροπή καλωσορίζει τη ε, γραμμή προπολογισμού για τις ε, ε, περιοχές με χαμηλό πληθυσμό γιατί ο παράγοντας αυτός θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει για την κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των κρατών μελών. Έχουμε θετική άποψη για το κοινοστρατηγικό πλαίσιο το Αγροτικό Ταμείο, το Ταμείο Ανάπτυξης Απέθρου και το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας θα πρέπει να ακολουθούν μια ενδυναμωμένη προσέγγιση και Φυσικά εδώ πρέπει να δούμε και ποιοι είναι οι στόχοι της στρατηγικής της Ευρώπης 2020. Θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Ταυτόχρονα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Πιστεύουμε ότι η πρόταση για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και για την ερωσιμότητα, δηλαδή τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να λάβει κάποιος στήριξη από την πολιτική συνοχής, βασικά έχουν καλές βάσεις ε, και οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια θα πρέπει να είναι σαφή και εύκολα να εφαρμοστούν. Διαφορετικά υπάρχει προφανής κίνδυνος ε, το σύστημα να καταστεί πολύπλοκο και να οδηγήσει σε μακρύς διαπραγματεύσεις ε, και σε αυξημένο διοικητικό άχθος. Αν πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες στον οικονομικό τομέα, τότε εγώ προσωπικά συμφωνώ με το κοινοβούλιο μας ότι θα προτιμούσαμε μείωση στην ε, γεωργική υποστήριξη, στην υποστήριξη στο γεωργικό τομέα ως ε, συντελεστή του πολιτικής συνοχής. Επίσης, υποστηρίζω την άποψη ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δίνεται έμφαση σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη, όπως ισχύει σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να περάσω στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, βγαίνει κυρία Φασίς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυρίλοφ. Ακούγοντας τους συναδέλφους ε, που τοποθετήθηκαν μέχρι τώρα, πίστευα ότι θα δεν μπορούσα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί η ουσία έχει εκφραστεί. Και μάλιστα, σε σχέση με που είπε ο προηγούμενος συνάδελφος από το Συνδικό Κοινοβούλιο, θέλω να υποστηρίξω τα όσα είπε. Φυσικά όλοι χρειαζόμαστε διαφανείς ε, συνθήκες, γιατί ακόμη και τα παλιά κρατημέλη έχουν δυσκολίες ε, με κάποιους όρους ε, και κάποιες προϋποθέσεις που τίθενται, καθώς όλο αυτό μας οδηγεί σε γραφειοκρατία. Όμως θα ήθελα να αναφέρω και ένα ευρύτερο ζήτημα γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα να έχουμε όλη την ίδια βούληση δράσης. Αυτό αφορά την ε, κατάσταση του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο σε σχέση με την πολιτική συνοχή. Κατά την άποψή μου, αυτό αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Και γιατί αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία και δεν νομίζω ότι αναμένεται ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει συμφωνία. Κάθε χώρα, τουλάχιστον κάποιες χώρες ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τίνουν απλώς ε, να εκριζωθεί αυτό που επιθυμούν ε, και αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Πραγματικά υπάρχει ένα σκιάχτρο πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό, αυτό συνίσταται στον εγωισμό των κρατών μελών. Αυτό δεν ισχύει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη έχουμε μία σαφή θέση και δεν ξέρω πόσο μακριά θα πάμε και σε αυτή τη μάχη. Και αν δούμε τη συνολική εικόνα, να σας πω ότι ε, ουσιαστικά ε, παλεύουμε για το σύνη πλήν 0,1% και φυσικά αυτό θα έχει αποτέλεσμα στην πολιτική συνοχή. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να δράσουμε από κοινού. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν ε, επενδύσεις στην ανάπτυξη από την πολιτική συνοχή με κάθε προϋπόθεση που θα μπορούσαμε να θέσουμε. Αλλά θα πρέπει να στραφούμε και στα Εθνικά Κοινοβούλια να ακουστεί η ανησυχία μας και θα πρέπει να επιμείνουμε. Δεν θα πρέπει ο κόσμος να καθορίζει την πολιτική συνοχή. Έχουμε κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον που θα πρέπει να καθορίζει την πολιτική συνοχή. Πρόσφατα, άκουσα από έναν ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπάρχει τουλάχιστον μία χώρα που ντρέπεται ακόμη και να μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάει απλώς για την ευρωπαϊκή αγορά και μόνο γι' αυτό. Και έχουμε δει και κάποιες ανησυχητικές δηλώσεις πρόσφατα ε, σε ό,τι αφορά τον ε, Βρετανό Πρωθυπουργό. Δεν εννοώ για την πολιτική συνοχή. Ξέρουμε όλοι πως έχει κατάσταση εκεί. Αλλά φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να έχουν κάποια παρέκκληση ό,τι αφορά την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Και ενώ μιλάμε για την ευρωπαϊκή αγορά, τι θα συνέβαινε αν κάποιες χώρες άρχιζαν να, να εφαρμόζουν ορισμένες παρκλήσεις, Τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύνολο. Και θέλω να κληρώσω με το εξής ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων των συναδέλφων στα Εθνικά Κοινοβούλια προκειμένου να προσδιορίσουμε την κατάλληλη πολιτική συνοχή. Είναι σημαντική αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά όλοι έχουμε κατανόηση για την οικονομική και χρηματομαστοποιητική κρίση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η πολιτική και κοινωνική κατάσταση σε κάθε χώρα. Αλλά όταν λέω ότι είναι κρίσιμη στιγμή, εννοώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι από κοινού προς αυτή την κατεύθυνση. Διαφορετικά δεν θα ωφεληθεί καμία χώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Και τώρα παρακαλώ να περάσουμε στην Πορτογαλία. Ασσαμπλέα τα Ρεπούμπλικα, ο κύριος Ονόριο Νόβου. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πραγματική ικανοποίησή μου να επιστρέφω στον οίκο αυτό κάποια έτη μετά από τις συζητήσεις τις οποίες ε, συμμετείχα στα τέλη της δεκαετίας του 90 σε άλλες αίθουσες, όχι σε αυτή εδώ. Και θα ήθελα εδώ να θέσω μια σειρά ερωτήσεων για να μας χρησιμεύσουν ως στοιχεία προβληματισμού είτε στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε ε, στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτη ερώτηση. Γιατί κάθε φορά στις πολιτικές συνοχής. Εισαγάγονται όλο ένα και περισσότερο κάποιοι στόχοι συνεργασίας με τρίτες χώρες που ε, σεβαστημένα, αλλά θα έπρεπε να χρηματοδετούνται με, μέσα από άλλη προέλευση και από άλλα κοινοτικά προγράμματα, ακόμη και στις περιπτώσεις που σε αυτές τις τρίτες χώρες, ε, αυτές οι τρίτες χώρες είναι όμορες χώρες, αλλά δεν είναι υποψήφιες προς 16 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Δεύτερη σκέψη γιατί ε, θέλουμε να επιβληθεί μια αποκλειστική ε, διάρθρωση των πολιτικών της συνοχής με τους στόχους ε, της Ευρώπης 2020, γιατί αρνούμαστε να σκεφτούμε με την ίδια βαρύτητα άλλα προβλήματα συνεργαζόμενοι στην ε, επίλυση άλλων συγκεκριμένων αναγκών διαφορετικών που θα μπορούσαν να υπάρχουν στο τάδε στο δίνα μέλος και ουσιαστικά θα ε, μπορούσε να είναι έτοιμα της στρατηγικής της Ευρώπης 2020, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία προηγήθηκε στρατηγικής Ευρώπη 2020, δεν είχε και πολλά αποτελέσματα. Τρίτη σκέψη, σε ένα γενικευμένο πλαίσιο κρίσης, ε, στο οποίο οι πολιτικές, επίσημες πολιτικές λιτότητας ε, ε, υλοποιούνται και ουσιαστικά δημιουργούν γενικευμένη ύφεση, και ε, επιδεινώνουν τις ασυμμετρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκαλούν ε, μεγέθυνση της ανεργίας και επιδεινώνουν την κατάσταση ε, στη ζωή πολλών Ευρωπαίων, κυρίως στις χώρες που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες και όπου υπάρχει εξωτερική παρέμβαση, γιατί οι πολιτικές συνοχές ε, θα πρέπει να ενισχύσουν την ερεσιμότητα, δηλαδή γιατί οι πολιτικές συνοχής ε, ουσιαστικά ρίχνουν λάδι στη φωτιά, αντί ε, να προσπαθήσουν να σβήσουν αυτή τη φωτιά. Τέταρτη σκέψη, γιατί σε ορισμένε περιπτώσει συγκεκριμένα κυρίως ε, για τις χώρες όπου ε, εφαρμόζεται ο μηχανισμός, που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό. Δεν ε, ξεκαθαρίζουμε σε ποια επίπεδα υπάρχει ορίμανση για τη χρημασία χρηματοδότηση σε όλες τις συνιστώσεις των προγραμμάτων. Τι περιμένουμε. Πέμπτη σκέψη, το θέμα της απλούστευσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός είναι ένας στόχος που πρέπει πάντα να επιτευχθεί. Πολύ ωραία. Ε, όμως ε, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που παρά τις ε, προσπάθειες απλούστευσης θα συνεχίσουν να υπάρχουν σε πολλά προγράμματα για ορισμένους πληθυσμούς και περιφέρειες και κυρίως σε ό,τι αφορά την ε, γεωργία σε οικογενειακό επίπεδο. Οι δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι πολλές φορές είναι ανυπέρβλητες και έκτο στοιχείο, έκτη σκέψη. Γίνεται πολλής λόγος ε, για την ε, υλοποίηση του κοινωτικού επιλογισμού και των πολιτικών συνοχής με έναν ισότιμο τρόπο. Επίσης γίνεται λόγος για ε, τις περικοπές που απαιτούνται από τις πολίτες. Τώρα εγώ θέλω να υπενθυμίσω δύο θέματα εδώ για να τα σκεφτείτε. Καταρχήν, στη δεκαετία του 90... Εγώ ήμουν μάρτυρας ότι ο Ζακ Ντελόρ ήθελε για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ε, ζητήσει 1,2% του ΕΠ για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό για 15 κράτη-μέλη. Δεύτερο σκέψη που θέλω να υπενθυμίσω, με μία ενιαία αγορά και με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, αγαπητοί συνάδελφοι, μήπως ε, και οι φορολογούμενοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι κύριοι δικαιούχοι των κοινοτικών πολιτικών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για τα σχολιά σας. Είναι μεγάλος ο αριθμός των ευρωβουλευτών. Οπότε θα αλλάξει λίγο η αναλογία. Θα έχουμε έναν εθνικό και έναν ευρωβουλευτή. Κύριε Σάμπρεχτ, κατάλαβα, Όλμπριχτ. Υπονοείται ότι πρέπει να είμαι σύντομο, Πρόεδρε. Ναι, ναι. Πέντε λεπτά νομίζω όμω ότι είναι πολλά, γιατί είσαστε συνηθισμένο στι μονόλεπτε παρεμβάσει. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Συναντιόμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή, όντως στιγμή κατά την οποία γίνεται ταυτόχρονα ο δημόσιος διάλογος για τα γενικά στοιχεία του κοινωτικού προϋπολογισμού, το πρώτο στοιχείο. Δεύτερον και στο παρόν κτίριο εξετάζεται, συζητείται η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια Ευρώπη με χαρακτηριστικά ευρωζώνης, ένα τμήμα προϋπολογισμού ειδικό, ένα τμήμα κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, ε, διαδικασιών. Συζητώντας λοιπόν την πολιτική συνοχής, θα πρέπει να έχουμε υπόψη όλοι, οι βουλευτές κάθε επίπεδου, ότι βρισκόμαστε, εγγραφόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο δημόσιο διάλογο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη μέθοδο που θα ε, μέσα από την οποία θα λειτουργήσει. Ε, εδώ λοιπόν η περιφερειακή πολιτική είναι η κοινοτική μέθοδος και εφόσον είναι η κοινοτική μέθοδος και αυτό είναι το κρίσιμο, απαιτείται μια σαφή σειρά κανόνων και η σύμπραξη των πάντων, των 27 δηλαδή κρατών μελών. Έτσι λοιπόν, υπεραμεινόμεθα της πολιτική συνοχής, αλλά δεν ζητάμε μόνο πιο πολλά χρήματα, ο μεν ή ο δε. Δεν μιλάμε μόνο για πιο πολλά χρήματα, μιλούμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η την κοινωνική μέθοδο, τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί για το μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό, αυτό το υπογραμμίζω γιατί θέλω να ε, υποσημειώσω ότι δεν πρόκειται για μια τεχνικού χαρακτήρα συζήτηση, αλλά για μια πολύ πιο ουσιαστική για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη κοινοτική μεθόδου. Αυτή ήταν μια πρώτη προκαταρκτική παρατήρηση. Για πιο συγκεκριμένα στοιχεία τώρα, θα ήθελα να υπογραμμίσω και να επισημάνω ότι το πρώτο στοιχείο που ανέφερε η Πρόεδρος αλλά και ο Επίτροπος οι συμβάσει εταιρική σχέση. Είναι, ε, εγγράφονται μέσα σε μια νέα φιλοσοφία. Δεν είναι τα παλιά, τα τετριμένα, τα γνωστά. Πρόκειται για μια νέα φιλοσοφία η οποία καταγράφει την αναγκαιότητα για συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων και αντιμετώπιση από κοινού των προβλημάτων της κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να, να αντιμετωπιστούν, να ξεπεραστούν οι διαφορέ μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Η Επιτροπή των Περιφερειών, εχθέ ε, στην αίθουσά μα εδώ, μίλησε για ένα κώδικα συμπεριφορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε επίση για ένα κώδικα συμπεριφορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά το αν είναι σκόπιμο να έχουμε ή όχι κώδικα συμπεριφορά, ενώ το Συμβούλιο τάσεται κατά ενό κώδικα συμπεριφορά, όχι αυτού καθεαυτού του κώδικα συμπεριφορά, αλλά κατά ενό συγκεκριμένου ε, μοντέλου κώδικα συμπεριφοράς για τις 27 χώρες μέλη. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους. Ποιοι είναι οι εταίροι, πώς θα συνεργαστούμε μαζί τους. Και πώς θα συνεργαστούμε όχι μόνο στη διατύπωση της σύμβασης, αλλά και σε όλη τη διάρκεια αυτή των 7 ετών, σε κάθε επίπεδο συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσει, με διάφορου εταίρου και ούτω καθεξής. Άρα θα είναι πολύ σημαντικό ο τρόπο με τον οποίο θα γίνει η σύλληψη, η περιγραφή και βέβαια θα χρειαστεί μια κοινή προσέγγιση, φαντάζομαι, μεταξύ των διαφόρων νομοθετικών οργάνων. Ε, Επίση, και μπορεί να φανεί τεχνική παρατήρηση, τεχνικού χαρακτήρα παρατήρηση, αλλά δεν είναι. Ε, το καθεστώ των συμβάσεων εταιρική σχέση. Και γιατί το λέγω αυτό, διότι η πρώτη βασική ιδέα ήταν η σύμβαση εταιρική σχέση να βασίζεται σε μια συμφωνία για το όλο σχέδιο, δηλαδή ποιο, με ποιο τρόπο, για ποιο λόγο, με ποιε ευθύνε, σε ποιο βαθμό. Εμεί ως Κοινοβούλιο προτείνουμε να προβούμε σε ένα πρώτο βήμα να καταλήξουμε σε μια πρώτη συμφωνία και μετά να προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Και η Επιτροπή πρότεινε τα λειτουργικά προγράμματα να συμβαδίσουν με την ε, σύμβαση εταιρική σχέση. Αυτή είναι η διαφορά, αλλά πολύ σημαντική διαφορά υπογραμμίζω, διότι είτε θα τα αντιμετωπίσουμε ως ε, ένα προκαταρκτικό τμήμα της διαδικασίας ή σε ένα πρώτο τμήμα πακέτου Αυτό νομίζω έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να το υπογραμμίσουμε γιατί έχουμε ξεκινήσει ήδη σε ορισμένα επίπεδα τη δουλειά. Επίσης, θεματολογικά τώρα. Συμφωνώ απολύτω με τον Επίτροπο Χάν ότι είναι καλύτερο από ένα μεγάλο μενού από το, να διαλέγουμε τρία πιάτα και όχι οχτώ μικρότερα μεζεδάκια. Το θέμα δεν είναι το νούμερο 8 ή 3, αλλά το περιεχόμενο βέβαια. Καλύτερα λοιπόν τα τρία πιάτα από τα 8. Η πρόταση όμω του Κοινοβουλίου πάνω απ' όλα είναι να μην αποφασίσουν οι Βρυξέλλε ποια θα είναι αυτά τα τρία πιάτα που θα βάλουμε στο μενού. Που θα βάλουμε μάλλον στο τραπέζι από το μενού. Να αφήσουμε αυτή την ευελιξία στι περιφέρειε. Και εμεί προτείνουμε να υπάρχει μια επιλογή, ένα περιθώριο κινήσεω, περισσότερη ευελιξία δηλαδή, για τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Χρειάζεται η συγκέντρωση, ναι, συμφωνώ απολύτω, αλλά αυτή δεν συνεπάγεται απουσία ευελιξίας στην ώρα που θα γίνει η επιλογή στην ε, κάθε περιοχή, στο κάθε, στον κάθε προορισμό. Τώρα, για να ολοκληρώσω τα πολιτικά δεδομένα, το πολιτικό πλαίσιο, Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το υπόλοιπο στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Θέλουμε συμβατικέ εταιρικέ σχέσεις, θέλουμε θεματική συγκέντρωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και πριν δώσω το λόγο στον προσεχή ομιλητή, θα πρέπει, ζητώντα συγγνώμη γιατί το παρέλειψα, να υπογραμμίσω ότι τον ε, κύριο Πρεσβευτή τον αντικατέστησε ως ο καταλληλότερος εκπρόσωπος του Συμβουλίου, ο Αντώνης Κωνσταντίνου, ο κύριος Αντώνης Κωνσταντίνου, ο οποίος ε, ε, προεδρεύει στην ομάδα εργασίας που διαπραγματεύεται και εξετάζει τις ε, ενδεχόμενες συμβιβαστικές λύσεις από πλευράς του Συμβουλίου και βέβαια θα είναι και ο συνομιλητής μας στους, τριμερείς, ε, στους άτυπους τριμερείς διαλόγους. Γι' αυτό σας καλώ, ανά πάσα στιγμή έχετε κάτι να σημειώσετε εκ μέρους είτε της Επιτροπής αλλά και του Συμβουλίου, να μας διακόψετε γιατί ασφαλώς θα ενδιαφέρονται στην αλήθεια να ακούσουν τις θέσεις σας. Ας ακούσουμε τώρα την Πολωνία, την Γερουσία, πρόεδρο τον κύριο Σέπιου, πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων. Συγγνώμη, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τα μικρόφωνα προς το παρόν. Σε ορισμένε περιπτώσει ε, οι δαπάνε ανακάτοικο είναι και ανώτερε, αλλά συνολικά η Πολωνία είναι μεταξύ των ε, ηγετών. Τουλάχιστον ε, αυτό θεωρούσα εγώ σήμερα. Η περίπτωση της Πολωνίας. Στην περίπτωση της Πολωνία. υπάρχει μια επιβεβαίωση τη αποτελεσματικότητας της πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πολωνία είναι η μόνη χώρα Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με την ε, διερμηνία προς τα γερμανικά. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Can you hear from the interpreters that there is any problem, or we can continue? No German. Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα το οποίο λύθηκε τεχνικό. Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε. Ξεραρχίζω λοιπόν, λέγοντας ότι η Πολωνία είναι καλό παράδειγμα για το πόσο αποτελεσματική, πόσο ουσιαστική μπορεί να είναι η Ευρωπαϊκή Συνοχή. Είναι το μόνο κράτος ε, που από το 2004 σημειώνει σταθερά ανάπτυξη. 1,7% το 2004, 2,5% φέτος ανάπτυξη χωρίς να υπολογίζονται τα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής. Φυσικά δεν θα είχαμε αυτήν την ανάπτυξη στην Πολωνία. Σημαντικό τώρα είναι το εξή. Έχουμε κάνει πολλές έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν ότι τα κονδύλια που απευθύνονται στην ε, Πολωνία, που εισφράττει η Πολωνία, έχουν ένα, παρουσιάζουν ένα φαινόμενο διάχυσης και ωφελούν τελικά και άλλα κράτη. Δεν πηγαίνουν δηλαδή τα οικονομικά ωφέλη μόνο στην ίδια την Πολωνία. Έχει μια προστιθέμενη αξία σημαντική αυτή η ευρωπαϊκή προσπάθεια. Αυτό προσπαθούμε πάντοτε να υπογραμμίζουμε ε, στις συνομιλίες μας και με τα άλλα κράτη μέσα από τη ε, διαδικασία που ονομάζουμε φίλοι της συνοχής. Εμείς από την Πολωνία υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερη οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική διαφοροποίηση έχει επίσης μεγάλη σημασία και πιστεύω ότι έτσι μπορούμε, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση ανά την Ευρώπη. Η εδαφική προσέγγιση είναι πολύ σημαντική, μια ολοκληρωμένη οριζόντια προσέγγιση που παρουσιάζει πιο πολλά πλέον εκτήματα. Τα κοινωνικά προγράμματα πλαισίου είναι πολύ σημαντικά, αλλά και τα λειτουργικά εθνικά προγράμματα. Οι συμβάσεις εταιρική σχέσης για μας έχουν επίσης πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει κατά την διαπραγμάτευση αυτών να εμπλέκονται όχι μόνο οι εθνικές αρχές αλλά και οι περιφερειακές, οι φορείς περιφερειακοί. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντική μια εξάντε συνεργασία εκ των προτέρων. Επίσης είμαστε πεπισμένοι ότι το 2017 και το, μέχρι το 2019 θα έχουμε μια θετική οικονομική αποτίμηση και ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαπραγματευτούν τα κράτη τους δείκτες για την αποτίμηση αυτήν ε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ανάπτυξη της, ε, των αστικών κέντρων επίσης ε, με συμβάσει εταιρική σχέσης μπορούμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των αστικών κέντρων ιδιαίτερως προσφέροντας επενδύσεις. Θα ήθελα βέβαια όμως να επισημάνω ότι υπάρχουν και επικρίσεις για ορισμένα σημεία. Το ζήτημα, η παραδείγματι, του φόρου προσθέμενης αξίας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα, ένα εκκρεμένο ζήτημα. δυσκολεύοντας ιδιαίτερα τις ε, ε μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο έργο τους. Και για να κλείσω, ένα πρόβλημα το οποίο θέλω να σας επισημάνω, το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe. Εδώ υπάρχουν δύο όψεις θα έλεγα ένα σημαντικό επιχείρημα κατά της πρότασης και άλλο ένα πολύ σημαντικό επίσης υπέρ. 10 δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να χορηγηθούν από το Ταμείο Συνοχής για την ε, δημιουργία ενός συμπληρωματικού συστήματος, αρκετά παρόμοιο με τον συνεπαγόμενο γραφειοκρατικό φόρτο και αυτό βέβαια θα είναι το ε, επιχείρημα κατά της ε, προαγωγής του μέσου αυτού. Αν δούμε ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ των προτάσεων για το Connecting Europe ε, και συγκεκριμένα σε σχέση με τα κράτη που ωφελούνται από αυτό, παράδειγμα την Πολωνία, μπορώ να υπογραμμίσω ότι προσπαθούμε, προσπαθούμε όλοι παραδείγματι να κατασκευάσουμε οδικού άξονε. Επιδιώκουμε όλοι την ε, διασύνδεση των πόλεων μας, αλλά τη διασύνδεση των κρατών μας με οδικούς άξονες δεν την έχουμε φροντίσει. Μπορεί να έχουμε πολύ πυκνό δίκτυο οδικό μέσα στα κράτη μας, αλλά η Τσεχία με την Αυστρία δεν έχουν καλή, ε, καλή οδική δικτύωση. Η Ουγγαρία με τη Ρουμανία, η, Σλοβακία με την Τσεχία. Δεν υπάρχουν καλές λοιπόν ε, ε, οδικές διασυνδέσεις. Όπω επίση, όχι μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το πρόβλημα θα το εντοπίσουμε και σε κράτη τη εγγύη γειτονία. Ουκρανία, Λευκορωσία, Τουρκία, ε, δεν έχουμε δίκτυα αυτοκινητοδρόμων όπως θα χρειαζόντουσαν. Ε, οι οδικοί άξονε που κατασκευάζονται συνήθω ε, κατασκευάζονται σε περιορισμένη έκταση, λίγα χιλιόμετρα μόνο και δεν επιλύουν τα προβλήματα. Και επίση δεν υπάρχει σωστή στόχοθέτηση και προτεραιότητε. Άρα λοιπόν, χωρίς μια επιπλέον δυνατότητα χρηματοδότηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέτοιου είδους ε, ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν. Ε, μέσα όπως το Connecting Europe μπορεί να αποτελέσουν ε, μια μεγάλη λύση, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πέραν των συνόρων για την διασύνδεση των περιφερειών μας και να επιτύχουν την επίτευξη, ή σε ένα βαθμό, την επίτευξη των στόχων που έχουμε προσδιορίσει. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι το, Ευρωπαϊκό, το Πολωνικό Κοινοβούλιο θεωρεί πως ρόλος του είναι να επιδιώκει και μια καλύτερη νομική βάση για την ε, συμμετοχή των διαφόρων οργανώσεων και φορέων ε, στην, ε, στην πολιτική της συνοχής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την άλλη λέει ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια μέσω της σύμβασης εταιρικής σχέσης με το multi-level governance. Αυτό μας υποχρεώνει να εξετάζουμε εάν μπορούν, τα, αν μπορούν οι ένομες τάξει μέσα στα κράτη-μέλη να προσφέρουν επαρκή νομική βάση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Όντω ε, η υπερσυνοριακή διακίνηση η οδική διασύνδεση είναι πολύ σημαντική, λέει η κυρία Χιούμπνερ, αλλά υπάρχει δυνατότητα μέσω τη ε, συνεργασία. Παρακαλώ. Ο κύριος Μάνκ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι και περιφερειάρχη στη Σλοβακία και ξέρετε ότι λόγω της κρίσης έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης του 20% γι' αυτό και χρειάστηκε να περιορίσουμε τις διοικητικές δαπάνες για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να υπάρξουν πόροι για νέες επενδύσεις, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ανάπτυξη. Θα σταματήσει ε, να λειτουργεί η ατομηχανή, αν θέλετε. Χάρη στην πολιτική συνοχή μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάποια έργα και μάλιστα σε κάποια κράτη-μέλη χωρίς συνοχή δεν θα υπήρχε καθόλου δημόσια επένδυση. Θα ήταν μηδενικό το στοιχείο αυτό. Επίσης είναι σημαντική συνοχή για την σύγκληση και την βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές στήριξης και για το δημόσιο τομέα, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως προείπε ο Πολωνός συνάδελφος, δεν ωφελούνται μόνο τα φτωχότερα κράτη από αυτή την πολιτική. Λόγω της ενέας αγοράς ωφελούνται και τα πλουσιότερα κράτη από την πολιτική αυτή, διότι παρέχουν τεχνογνωσία, προϊόντα και υπηρεσίες στις άλλες χώρες. Θέλω λοιπόν να σας υπενθυμίσω την κοινή διακήρυξη, την κοινή δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων 15 κρατών μελών φίλη συνοχή στη, Βρα... στη Βρατισλάβα την προηγούμενη εβδομάδα 11 νέοι, 3 παλιοί και η Κροατία ήταν παρόντε εκεί. Η Κροατία σύντομα θα γίνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν παρόν ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι του είπαν ότι η πολιτική συνοχή είναι ένα βασικότατο επενδυτικό εργαλείο για όλα τα κράτη-μέλη. Εάν λοιπόν μειωθεί η χρηματοδότηση στον τομέα αυτό, δεν πρόκειται να επιτύχουμε του στόχου του Συμβουλίου το οποίο αναβάθμισε τις φιλοδοξίες του σύντομα ανοιοθετώντας ε, τα συμπεράσματά του. Δεν θα πετύχουμε τους στόχους ε, της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Όπως είπαν και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, δεν πρέπει να περιοριστούν οι πόροι της τη συνοχή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να πω, ότι κατά πλειοψηφία τάσεται υπέρ της ε, αυξήσεως των πόρων της συνοχής. Αγαπητοί συνάδελφοι, χρειαζόμαστε όμω τη στήριξη και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο, σε σχέση με τον Ιρλανδό συνάδελφο, που είπε ότι είναι μια επιτυχημένη ιστορία η Ιρλανδία σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχή. Πράγματι, ήμουν πριν από κάποια χρόνια στην Ιρλανδία, γιατί ήμουν εισηγητή για τον κοινοτικό προπολογισμό και είχα συνομιλίε τότε με τον ε, Ιρλανδό Υπουργό Οικονομικών. Γιατί το αναφέρω, γιατί τίθενται δύο διαφορετικά θέματα εδώ. Εγώ ως περιφερειάρχη στην ε, Σλοβακία σκέφτομαι ότι και εγώ θα ήθελα να μπορέσω να αξιοποιήσω στον το περισσότερα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής στην δική μου περιφέρεια. Έχουμε όμως το παράδειγμα της Ιρλανδίας που έκανε κεντρικά, συγκέντρωσε τους πόρους, αν και μικρή χώρα, συγκέντρωσε όμως τους πόρους και τελικά κατάφερε να πετύχει το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφηση αυτών των κονδύλων στην Ευρώπη. Οι εταιρικέ σχέσεις λοιπόν είναι το σημείο κλειδί εδώ. Εταιρικέ σχέσεις μεταξύ πόλεων, κομοπόλεων, χωριών κτλ. ώστε να συμφωνηθεί μεταξύ τους ποια είναι η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση αυτών των κονδύλων. Να περάσουμε τώρα στην Ισπανία, λέει η Πρόεδρος από τη Βουλή. Ο κύριος Μανουήλ Γκονθάλη θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ένα θερμό χαιρετισμό σας απευθύνω από την Ισπανία. Μιλάμε για την πολιτική συνοχή. Η Ισπανία έχει εμπειρία όπως άλλες περιφέρειες, όπως άλλες χώρες για το πόσο θετικό αντίκτυπο είχε η πολιτική συνοχή. Ήταν αποτελεσματική, ωφέλησε πολλές περιφέρειες, άρα και πολλούς ανθρώπους, πολλούς συμπολίτε μας. Δεν θα μιλήσουμε για την κρίση. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης ε, ε, πληττόμεθα από μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση. Η υπόλοιπη Ευρώπη όμως μπορεί να κάνει πολλά για να βοηθήσει για να δείξει την αλληλεγγύη τη σε όλε τι χώρε. Και εγώ βέβαια μιλώ εδώ εξ ονόματο τη Ισπανία. πάνω περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να υπάρξει σύγκληση, αλληλεγγύη μεταξύ περιφερειών. Στην Ισπανία έχουμε κάποιες, αρκετές θα έλεγα, περιφέρειες, κατηγοριοποίηση στις λεγόμενες περιφέρειες σε μεταβατική περίοδο. Τώρα λοιπόν που σκεφτόμαστε την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είναι πιο απαραίτητο από ποτέ οι χώρες εκείνες που θεωρούν οι ίδιες ότι συνεισφέρουν ε, καθαρά στον πεπλισμό, αλλά εγώ νομίζω ότι όλοι συνεισφέρουμε τέλος πάντων, αλλά οι χώρες που θεωρούν ότι είναι καθαροί εισφορείς επιμένω ότι αυτές οι χώρες πρέπει να δείξουν ακόμα μεγαλύτερη αλληλεγγύη, διότι η ανάπτυξη χωρών όπως η Ισπανία συνεπάγεται ανάπτυξη για όλη την Ευρώπη. Εάν θέλουμε λοιπόν με περισσότερη Ευρώπη, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερη Ευρώπη, αυτό θα το πετύχουμε αν είμαστε αλληλέγγυοι. Επιμένω στη λέξη αλληλεγγύη. Και επειδή πολλέ περιφέρειες ε, στην Ισπανία είναι σε μεταβατική περίοδο, χρειάζονται περισσότερο από ποτέ αυτή την πολιτική συνοχή, τα ταμεία, τα κονδύλια συνοχή. Όπω πολύ καλά είπε ο Επιτρόπος και συμφωνώ μαζί του, ο δημοσιονομικό αυτό ο αυτέ αυτές οι πολυετής προοπτικέ μέχρι το 2020 δηλαδή, θα δώσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην Ισπανία, όχι στην Ευρώπη. Φυσικά και στους Ισπανούς βέβαια, αλλά στους Ευρωπαίους εν γέννη, διότι αν υπάρχει μια οικονομική προοπτική ε, που σημαίνει ότι οθούμε και βελτιώνουμε την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη, τελικά τι κάνουμε, βοηθάμε την Ευρώπη. Βοηθάμε τις υπόλοιπες χώρες, τις περιφέρειες και κυρίως τους ανθρώπους, γιατί γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Άρα περισσότερη συναματοδότηση, περισσότερη αλληλεγγύη, ενίσχυση των πολιτικών συνοχής των περιφερειών στην προκειμένη περίπτωση της Ισπανίας, αλλά και όλων των άλλων χωρών που χρειάζονται αυτή τη στήριξη. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much, ε, Madam Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ τους ε, μιλητές για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι το θέμα του προπολογισμού είναι το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή και το πολιτισμικό συνομικό πλαίσιο. Άκουσα τι είπαν οι ομιλητέ και τον Επίτροπο Χάν. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε κάθετοι επ' αυτού. Δεν θα πρέπει να μιλάμε αυτή τη στιγμή για μειωμένο προπολογισμό. Και δεύτερον, συμφωνώ με τον Ισπανό συνάδελφο που αναφέρθηκε στο ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στους φορολογουμένους και στους δικαιούχους. Όλοι είμαστε φορολογούμενοι και όλοι είμαστε δικαιούχοι. Και νομίζω ότι δεν θα έβλεπτε αν ε, οι χώρες ε, που ε, κάνουν πολύ φασαρία ότι είναι καθαροί συνεισφέροντες να τονίσουν τι σε αυτές την προσθεμένη αξία του να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενιαία αγορά και στην ενιαία αγορά, αλλά και σε επίπεδο περιφερειών σε αυτά τα κράτη-μέλη, τα οποία πάρα πολύ έχουν ωφεληθεί από το Ταμείο Συνεχής ε, και από άλλα κονδύλια τα τελευταία χρόνια. Όπως ε, είπε και ο συνάδελφος από την Ιρλανδία, η Ιρλανδία έχει ωφεληθεί τα μάλα από την Ευρώπη, από την πολιτική συνοχή στα χρόνια όταν εμείς ε, ε, ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμασταν στο 58% του μέσου όρου του ΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτάσαμε στο 124% και τώρα επαναχωρήσαμε λόγω των προβλημάτων των τραπεζών και των υπερβολικών δαπανών και όλα αυτά μας οδήγησαν ε, στα μέτρα λιτότητας, όμως ε, η βασική υποδομή που συστάθηκε από την πολιτική συνοχή ε, στην Ιρλανδία παραμένει. Και αυτό ωφελεί πάρα πολύ και όταν θα επανέλθουμε σε καλύτερη κατάσταση θα μας βοηθήσει. Και όπως υπόθηκε, σε όλη τη χώρα υπήρξαν ωφέλη, άνοιξαν διάφορες οδικοί οδοί ε, βάσει της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ε, και πρέπει να κάνουμε περισσότερα προς αυτήν την κατεύθυνση για να δουν οι πολίτες τα ωφέλη. Γιατί η αρνητικότητα μας ε, καταποντίζει. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε κάθε συζήτηση και έχουμε υποχρέωση να υπερασπίσουμε την πολιτική συνοχής, να υπερασπίσουμε τον προπολογισμό και σε αυτή τη χρονική στιγμή, ούτε σε καμία χρονική στιγμή, δεν θέλω να λέμε θα πρέπει να διατηρήσουμε τον προπολογισμό ε, για την πολιτική συνοχή. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για καμία περικοπή αυτή τη στιγμή. Έχουμε καλέ πολιτικέ, η Ευρώπη, Ευρώπη σημαίνει ελληνική. Όλους τους ωφελεί. Έτσι λοιπόν ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο 1,3 ε, που ζητάει η Κομισιόν στον προπολογισμό έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε για να βγούμε από την ύφεση. Μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη και μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής ε, της Ευρώπης 2020 και των 7 θεματικών πρωτοβουλειών. Ε, εμείς δεν θέλουμε να αποτύχουμε όπως αποτύχαμε στη στρατηγική της Λισαβόνας και η συνοχή θα διαδραματίσει πολύ μεγάλο ρόλο στο να διασφαλίσει ότι δεν θα αποτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ Σαμ. Τώρα θέλω να καλέσω την κυρία Στέλλα Δημητρίου να πάρει το λόγο από την Κύπρο. Κυρία Πρόεδρε, ε, αρχικά θα ήθελα πριν από στην ουσία να πω ότι ε, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση στην πολύ πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης στην Κύπρο στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πραγματοποιήθηκε μια πολύ ωφέλιμη συζήτηση και υπογραμμίστηκε σε αυτήν την κοινή συνεδρία που ήταν από δική μας πλευράς οι Επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αλλά και η Επιτροπή Εσωτερικών. Ε, υπογραμμίσαμε και ανταλλάξαμε έτσι, απόψεις και θέσεις πάνω στην πολιτική της κοινωνικής συνοχής. Υπογραμμίζω ιδιαίτερα ότι είναι ωφέλιμες αυτές οι επισκέψεις και η ανταλλαγή απόψεων ή στι χώρε μας ή στα εθνικά μα κοινοβούλια που μα δίνεται ευκαιρία να γνωριστούμε και από κοντά. Ε, παρόλο που ο, ο κύριος πρέσβης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, μίλησε εκτενέστερα για το θέμα που συζητούμε σήμερα και εγώ με τη σειρά μου θέλω να υπογραμμίσω κάποια ε, ιδιαίτερα θέματα και να θέσω τις ε, απόψεις μας περί αυτών το, νομικό, το νέο πλαίσιο νομοθετικών μέτρων που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2011 και αφορά το διάστημα 2014 μέχρι 2020 θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των κυβερνήσεων αφού περιέχει απλουστευμένες διαδικασίες οι οποίες εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο έχοντας υπόψη τα πολύ επίγοντα ζητήματα που φιλοδοξούμε να επιλύσουμε με τη σχετική πολιτική. Μέσα από αυτές τις κοινέ πρόνοιες πιστεύω ότι θα επιτευχθεί μια πολύ διευρυμένη πρόθεση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, των έργων υποδομής αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών. Θέλω να πω επίσης ότι ε, οι προτάσεις για το νομοθετικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής μέχρι το 2020 δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την Κύπρο. Η Κύπρος έχει καταταχθεί στην κατηγορία των πιο ανεπτυγμένων περιφερειών με κριτήριο το κατακεφαλή ακαθαρίστο εθνικό προϊόν που αυτό εξυπακούει το 90% του μέσου όρου των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και με δεδομένων αυτήν την κατάταξη η Κύπρος λαμβάνει μειωμένη κατανομή κοινοτικών πόρων, σχεδόν το 1 τρίτο των πόρων της τρέχουσας περίοδου σε συνδυασμό με αυξημένους περιορισμούς ως προς τη χρήση των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για τις περιοχές αυτές μειώνονται από το 85% σε 50%. Η επικέντρωση των παρεμβάσεων σε περιορισμένο αριθμό θεματικών προτεραιοτήτων των ταμείων, ιδιαίτερα στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες που προτείνει η Επιτροπή, δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές περιφερειών των κρατών με συγκεκριμένα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και φυσικά μειονεκτήματα, όπως είναι τα νησιά για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης που λέει ότι σε νησιώτικες περιοχές μπορεί να περιλαμβάνει και νησιά κράτη ε, εφόσον ικανοποιούν τα αναγκαία κριτήρια. Να πω επίσης ότι ε, με το δίκτυο ασφαλείας η Κύπρος ε, εξακολουθεί να μην διασφαλίζει το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό που χρειάζεται η χώρα ώστε να ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές της ανάγκες και προοπτικές. Παρόλο που υπάρχει αυτή η αναφορά στην ειδική περίπτωση των νησιώτικων περιφερειών στο διαπραγματευτικό πλαίσιο, ε, δεν διευκρινίζεται πώς θα παρέχεται και με ποιον τρόπο θα λαμβάνονται υπόψη αυτές οι ειδικέ περιπτώσεις. Η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής του 2007-2013 καταδεικνύει ότι θα ήταν ωφέλιμη η ενεργότερη και από τα αρχικά στάδια συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και των κυβερνήσεων ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει έγκαιρα και έγκυρα τα σωστά μηνύματα για τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των επιμέρους περιφερειών. Η όλη φιλοσοφία της πολιτικής συνοχής διαπνέεται από την ανάγκη για καταπολέμηση των ανισοτήτων και του χάσματος ανάμεσα στις περιφέρειες της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτόν τον λόγο απαιτείται η προδιαβούλευση μεταξύ των εν φορέων για ορθότερα και πιο στοχευμένα αποτελέσματα. Η επιτυχής διαχείριση της πολιτικής συνοχής αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει σαν στόχο την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης των νομοθετικών προτάσεων που θα πλαισιώνουν την πολιτική συνοχή της περίοδου 2014-2020. Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στηρίζει οποιαδήποτε προσπάθεια η οποία στοχεύει στην προώθηση ανθρωποκεντρικών πολιτικών αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθημερινότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Γι' αυτό θα σταθεί αρρωγός για την έγκαιρη ή δυνατόν ολοκλήρωση της σχετικής διαπραγμάτευσης. Και πριν να κλείσω, θέλω να υπογραμμίσω ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει ετοιμάσει και αποστείλει αναθεωρημένο κείμενο του διαπραγματευτικού πλαισίου που ε, αναθεωρεί και περιλαμβάνει πρόνοια για ενδεχόμενη αύξηση του δικτύου ασφαλείας για τους πόρους που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες και να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτός ο θεσμοθετημένος διάλογος ε, με τα κοινοβούλια λαμβάνει χώρα και μάλιστα πάρα πολύ επίκαιρα γιατί ε, είναι επίκαιρο όχι μόνο βέβαια για την πολιτική συνοχή αλλά και για την Ευρώπη το να συζητάμε αυτά τα θέματα. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόσο, έδωσε μια πάρα πολύ αξιοσμένη ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είπε ότι πρέπει να προωθήσουμε το ομοσπονδιακό μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ στηρίζω πλήρω αυτή την ιδέα το να ε, καθιδρύσουμε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ομοσπονδιακό σύστημα. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι και τα εθνικά κοινοβούλια, τα κράτη-μέλη θα μεταφέρουν ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι εθνικής κυριαρχίας στις Βρυξέλλες και στο, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κατά την ταπεινή όμως ε, άποψή μου, το ομοσπονδιακό μοντέλο μπορεί να καταστεί βιώσιμο μόνο αν συνοδεύεται από αλληλεγγύη και η πολιτική συνοχής είναι ακριβώς ε, ε, το εργαλείο που μπορεί να αντιμετωπίσει ανισότητες ε, εσωτερικά στα κράτη-μέλη αλλά και μεταξύ κρατών μέλων. Και στην πράξη δείχνει ε, ότι πραγματικά την αλληλεγγύη την εννοούμε. Δεν είναι μόνο στα λόγια αλλά γίνεται και πράξη. Είμαι πεπισμένος ότι η ιδέα περιστολής ε, των δαπανών για την πολιτική συνοχή θα υπονομεύσει οποιαδήποτε δυνατότητα να προοδεύσουμε και πρέπει να το δεχθούμε. Με τα υφιστάμενα εργαλεία και μέσα η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει. Μην ξεχνάμε φίλοι όμως το εξής. Το 2014 έχουμε ευρωεκλογές και μας αφορά όλους τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη, τα εθνικά κοινοβούλια, τα εθνικά κόμματα. Πώς θα πλασάρουμε ε, το ομοσπονδιακό μοντέλο την Ευρώπη ε, το 2014. Γιατί τα κόμματα που θα κατέβουν στι εκλογές ε, το 2014 μπορεί να έχουν και το δικό τους υποψήφιο τον πρόεδρο της Κομισιόν. Πώς μπορούμε λοιπόν και στους Ευρωπαίους πολίτες να κάνουμε να σπαστούν την ιδέα αυτή και να εργαστεί το, το Κοινοβούλιο για τις νέες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν, πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά, όταν κάποια κράτη-μέλη λένε ας έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο για τον προβλησμό της Ευρωζώνης. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να πετύχεις καλύτερα να υπονομεύσεις αυτή την προσπάθεια για μια καλύτερη Ευρώπη και για περισσότερη Ευρώπη, κάτι που χρειαζόμαστε όλοι. Και ολοκληρώνοντας αυτή τη γενική πολιτική τοποθέτησή μου, μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Αν γίνω κοινικό, μπορώ να πω ότι η μόνη δυνατότητα τα 27 κράτη-μέλη όσα άλλα στο μέλλον προσχωρήσουν, Κροατία που είναι σίγουρη και όποια άλλη. Τα 27 λοιπόν και παραπάνω όσα κράτη-μέλη μπορούμε να γίνουμε ένας παγκόσμιος πρωταγωνιστής μόνο εάν επανέλθουμε στα εθνικά συστήματα με τα εθνικά κράτη-μέλη. Αν επανέλθουμε θα είναι και η Γερμανία ένας νάνος μπροστά στην Κίνα τότε. Πώς ε, θα συγκριθεί δε με μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα και τα λοιπά, φανταστείτε η Μάλτα, η Σλοβακία και τα λοιπά. Αν θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει να έχουμε την απαιτούμενη μόχλευση και την πρόοδο που θέλουμε, αλλιώς θα υπονομεύσουμε την Ευρώπη. Πρέπει να επιλέξουμε το ένα το άλλο. Και είμαι βέβαιο ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια θα εργαστούν για μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση το όνομα τη αλληλεγγύη, γιατί αυτή είναι η μόνη αξία πάνω στην οποία μπορούμε να θεμελιώσουμε την Ευρώπη. Τώρα, έρχομαι στην άλλη όψη του νομίσματο. Και θα μιλήσω και ρουμανικά, γιατί αφορά πιο πολύ τα εσωτερικά ζητήματα της, ε, που αντιμετωπίζει σήμερα η Ρουμανία. και συγκεκριμένα αφορά τη θεσμική και διοικητική ικανότητα. Όλα τα έγγραφα που εκπώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκινώντας από τους γενικούς κανονισμούς και φτάνοντας σε ειδικού κανονισμούς, είτε για τα ταμεία, είτε για το μέσο συνέντες στην Ευρώπη, όλες οι πρωτοβουλίες αυτές Έχω ψύχωση με τη φράση πρέπει να αυξήσουμε τη διοικητική και θεσμική δυνατότητα και ικανότητα αν θέλουμε η νέα πολιτική συνοχή να δώσει αυτά αποτελέσματα για τις κοινότητες, για τις περιφέρειες, για τα κράτη-μέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι προφανές ότι θα επιτελέσει το καθήκον του. Έχουμε τη στήριξη της Κομισιόν και νομίζω ότι καταφέραμε να ε, απλουστεύσουμε τα έγγραφα. Αναλύστε όμως περισσότερο τα έγγραφα αυτά για να δείτε. Μιλάμε για νέους μηχανισμούς, για νέους θεσμούς. Όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν, να είναι επιχειρησιακά από 1η Ιανουαρίου του 2014. Υπάρχουν πέντε ταμεία που διέπονται από τους ίδιους κανονισμούς για να έχουμε αυτή την πολυεπίπεδη προσέγγιση, πολυταμιακή προσέγγιση. Και για να έχουμε τα αποτελέσματα που αναμένουμε από την πολιτική συνοχή, πρέπει αυτά ε, τα όργανα, αυτοί οι φορεί να είναι επιχειρησιακοί από 1η Πρώτου 2014. Πρέπει λοιπόν να ασκηθεί πίεση και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γνωρίζω ότι κάποιες χώρες ε, κάνουν καταπληκτική δουλειά. Η Πολωνία είναι το αγαπημένο παράδειγμα και είμαι πολύ περήφανος που μια πρώην κομμουνιστική χώρα έχει γίνει πηγή έμπνευση για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Πρέπει όμως τα Εθνικά Κοινοβούλια να επανεξετάσουν την κατάσταση και να φτιάξουν μια λίστα που θα περιλαμβάνει το τι δεν πήγε καλά, τι λείπει ε, σε ό,τι αφορά τη διοικητική ικανότητα των κρατών, τι πρέπει να διορθωθεί τάχιστα από νομικής και θεσμικής πλευράς ώστε όταν έλθει 1η Ιανουαρίου του 2014 να είμαστε έτοιμοι και να μπορούμε να πούμε ορίστε, να η νέα πολιτική συνοχής που μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να φέρει καρπούς, να δώσει θετικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος και συγγνώμη που μιλάω έτσι λίγο μερκαντιλιστικά, ε, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να πουλήσεις, να πλασάρεις στην Ευρώπη από το να προωθήσεις την πολιτική συνοχής να διαφημίσει την πολιτική συνοχή στου δρόμους, στι πόλεις, στα χωριά. Αυτό αποτελεί υποχρέωση. Αλλά είναι και κυρίαρχο δικαίωμα ταυτόχρονα των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δηλαδή, να φροντίσουν το τεράστιο αυτό δυναμικό, αναπτυξιακό δυναμικό, δηλαδή η θεσμική και διοικητική ικανότητα, θα βελτιωθεί ώστε αργότερα να μπορούμε να μιλάμε για την επιτυχημένη εφαρμογή του νέου πλαισίου συνοχής. Ευχαριστώ, Πρόεδρος επειδή ο, ο κύριος Αντώνης Κωνσταντίνου πρέπει να μας εγκαταλείψει σύντομα, θα του δώσω τώρα το λόγο εκ μέρους τη Προεδρίας για δύο-τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την οργάνωση αυτής της συνάντησης. Άκουσα με μεγάλη ικανοποίηση τις απόψεις των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια Καταρχήν, ε, η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στο εθνικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν έχει παρέμβει στη διαδικασία αυτή αλλά υπάρχουν ε, κάποια εργαλεία όπως έλεγχος επικουρικότητας και νομίζω ότι είναι σημαντικό τα εθνικά κοινοβουλία να συμμετέχουν σε αυτή την πολύ σημαντική πολιτική. Η πολιτική της συνοχής είναι σημαντικό να έχει συγκεκριμένους στόχους για την επίτευξη της συνοχής των περιφερειών των κρατών μελών. Όμως τώρα πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που τα νέα στοιχεία της νέας πολιτικής ε, συνοχής θα μας οδηγήσουν στο να μετακινηθούμε από την πολιτική αυτή, ε, στο να την καταστήσουμε σε ένα κύριο αναπτυξιακό μέσιο της Ένωσης. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά η προσωπική μου φιλοδοξία και όνειρο είναι να δω την πολιτική συνοχή, να αποτελεί την κύρια αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Και νομίζω ότι υπάρχουν ε, ορισμένα βήματα, πέρα από άκουσα σήμερα, άκουσα πολλούς από τους ομιλητές να αναφέρονται σε κονδύλια και σε πόρους. Φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ζωτικό. Ω εκπρόσωπο Προεδρία, δεν μπορώ να σχολιάσω ιδιαίτερα τι συζητήσει που κάνουμε για το πολιτέ πλαίσιο, αλλά μπορώ να σα διαβεβαιώσω για το εξή. Η Προεδρία θα διασφαλίσει ότι η κοινοτική μέθοδο θα ακολουθηθεί στη, στο σύνολο των συζητήσεων και ότι η η πολιτική συνοχή ε, θα διέπεται από ορισμένα κριτήρια. Τα έχει δηλώσει αυτά η Προεδρία, ποια, δηλαδή ποια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για να καθοριστούν τα ποσά για κάθε, πολιτικής, για κάθε πολιτική. Και η πολιτική συνοχή είναι μια σημαντική πολιτική, δυνάμει και των συνθήκων και ε, αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε και τι ισχύει και στην προηγούμενη περίοδο. Όμως δεν μπορώ να πω πολλά για τη χρηματοδότηση γιατί οι συζητήσεις ε, είναι σε εξέλιξη, αλλά μπορώ να σας πω κάποια λόγια για το περιεχόμενο της πολιτικής. Ε, τα τρία όργανα έχουν μια κοινή ε, κατανόηση, υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά υπάρχει κοινή κατανόηση σε σχέση με τη νέα προσέγγιση της πολιτικής συνοχής, σε σχέση με τα νέα στοιχεία αυτής. Και νομίζω ότι και οι τριστασμοί συμφωνούν επί τη στρατηγική προσέγγιση. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της πολιτικής, προκειμένου να συνδυάσουμε όλα αυτά τα ταμεία και όλα αυτά τα ταμεία ε, να εργαστούν σε συνέργεια. Και νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Φυσικά έχουμε και ένα δεύτερο θέμα, τη θεματική συγκέντρωση, πολιτική συνοχή, όπω υπόθηκε και από τον Επίτροπο και άλλου ομιλητέ, θα πρέπει να συνεισφέρει στην επιτεύξη των στόχων τη Ευρώπη 2020, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε κράτος μέλος και κάθε περιφέρεια λαμβανομένων υπόψη και των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων. Γι' αυτό το Συμβούλιο πιστεύει ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποια ευελιξία. Και άκουσα σήμερα να λέγεται ότι ένα μέγεθος δεν κάνει για όλους. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι η ευελιξία θα μπορούσε να συνεπάρξει με την ολοκληρωμένη προσέγγιση και αυτές είναι οι δύο όψεις νομίσματος της αηφόρου ανάπτυξης. Και θα ολοκληρώσω με το εξής το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και οι διαπραγματεύσεις ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικές. Η Προεδρία έβαλε την δυνατά της ενεργαστή προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ο πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα κάνει επίσης μια προσπάθεια για να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις μέχρι τον Νοέμβριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να στείλω αυτό το μήνυμα σε όλα τα μέρη ότι για την πολιτική συνοχής μία αργή συμφωνία, δηλαδή μετά τα τέλη του 2012, θα είναι καταστροφική. Γιατί αν έχουμε μία καθυστερημένη συμφωνία, ξέρετε ε, πόσος χρόνος χρειάζεται για να προετοιμαστούν τα προγράμματα Όλοι οι αρμόδιοι το ξέρουν και θα πρέπει να υιοθετηθούν και οι κανονισμοί μετά τη Συμφωνία για το Πολιτέ Δημοσιονομικό και προηγούμενε περιόδου. Ξέρουμε ότι χρειάζονται ένα με δύο έτη για την προετοιμασία. Επομένω, δεν μιλάμε για μια πολιτική όπω οι άλλε, όπου έχουμε μια αιτήσια πληρωμή ε, και τα εισοδήματα κτλ. Επομένω, το Κοινοβούλιο αλλά και όλοι οι θεσμοί των ε, κρατών μελών πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το χρονοδιάγραμμα και η Προεδρία έβαλε τη δυνατά τη προς την κατεύθυνση αυτή. Κάτι ακόμη τώρα, γιατί περιμένουμε για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Προεδρία έχει θέσει ένα πολιτικό στόχο στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων ε, του πακέτου της συνοχής. Δηλαδή να ολοκληρωθεί ο διοργανικός διάλογος μεταξύ των τριών οργάνων σε μια πτυχή που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους πολίτες και για τα κράτη-μέλη, τον προγραμματισμό όλα τα κράτη-μέλη, όλες οι περιφέρειες ε, και όλοι οι αρμόδιοι γνωρίζουν ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού, ποιο είναι το πλαίσιο που θα αρχίσουν να προετοιμάζουν. Ελπίζω λοιπόν ότι και τα άλλα δύο όργανα και είμαι σίγουρος ότι ήδη και οι υπόλοιποι εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν ελπίζω ότι πριν τα τέλη του έτους να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αν δεν καταρθώσουμε, μάλλον να ολοκληρώσουμε το σύνολο του κανονισμού, τουλάχιστον να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την κοινή συνεννόηση επί αυτών των σημαντικών πτυχών του προγραμματισμού. Έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να προετοιμαστούν όσο το, δυνατόν συντομότερα στην περίπτωση που δεν έχουμε συμφωνήσει από του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σα και θα παρακολουθούμε στενά το έργο σα. Σα ευχαριστώ. Καλό τώρα τον κύριο Στέφαν Μάιερ, εκπρόσωπο της Μπούντες, θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή την διακοινοβουλευτική εκδήλωση, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη και κυρίως το γεγονός ότι μέσα από τον τριμερή διάλογο, όπως είπαν οι περισσότεροι από τους παρεμβαίνοντες, διαμορφώνεται η διαρθρωτική πολιτική. Ιδιαίτερα σημασία έχει για να έχουμε μια καλή περιφερειακή πολιτική όπως τη ζητούμε στο, Ευρωπαϊκό, στο Γερμανικό Κοινοβούλιο να, να επιδιώκουμε μέσα από τη στρατηγική αυτή τους στόχους της Ευρώπης 2020. Προς αυτήν θα πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι και στην προσεχή περίοδο νομίζω ότι θα ε, καταστεί αυτό ακόμη πιο σαφές, ενώ βέβαια και των προσφατών εξελίξεων και της εμπειρίας που έχουμε συλλέξει στην Ευρώπη, ότι θα χρειαστεί να δώσουμε λύσεις και για την ανεργία ιδιαίτερως ε, μέσα από την περιφερειακή πολιτική, μέσα από την τερθωτική πολιτική. Ιδιαίτερα θα πρέπει να καταστήσω σαφές ότι με τις ε, πρόσφατες ε, εμπειρίες που έχουμε το μέλλον θα εξαρτηθεί ιδιαίτερα από την δυνατότητα να τηρήσουμε τις προϋποθέσεις του προϋπολογισμού, τη δημοσιονομική δηλαδή ε, υγιή δημοσιονομικά, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και να ε, προαθήσουμε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με βάση ιδιαίτερα την καινοτομία. Για να προσδιοριστεί όμως η καινοτομία θα πρέπει να αφήσουμε πιστεύω ένα περιθώριο ευρύτερο επιλογών και να μιλήσουμε για την πραγματικά παραγωγική ανταγωνιστικότητα. Φερρυπίν ε, για μετάθεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό, πιο παραγωγικό. Και επίσης για το μέλλον. Στο πλαίσιο της, περιφερειακής, ε, της πολιτικής συνοχής και της αγροτικής πολιτικής θα πρέπει να εμπλακούν όλες, νομίζω, οι περιφέρειες ε, και επισημαίνω ότι κατά την άποψή μας με το να αποδυναμώνονται οι πιο ισχυρές περιφέρειες δεν ενισχύονται απαραίτητα οι πιο αδύναμες. Έτσι λοιπόν πρέπει σε ένα προσεχές δίκτυο ε, στήριξης να συμπεριλαμβάνονται όλες οι περιφέρειες. Πολύ σημαντικό είναι, όπως άλλωστε ήδη έχει προβλεφθεί, να ενισχυθεί η, η διαπεριφερειακή συνεργασία πράγμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταστήσουμε σαφές στον πολίτη πόση μεγάλη αξία προσφέρει η Ευρώπη. Αυτή η διαπεριφερειακή λοιπόν συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο της εδαφικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα θα για μένα και άλλωστε θα πρέπει με επικριτικό βλέμμα να το εξετάσουμε, να δούμε αν στην προσεχή περίοδο στήριξης 14-20 έχει σκοπιμότητα να ζητηθεί η, πλήρω, η πληρώση και των τεσσάρων κριτηρίων που προβλέπονταν. Γιατί μέχρι τώρα προβλεπόταν ε, τα δύο κράτη που συνεργάζονταν να πληρούν δύο μόνο κριτήρια. Τώρα προτείνεται να διπλασιστεί αυτή η αιρεσιμότητα, να είναι πιο αυστηρά, ε, δηλαδή προδιαγραφές και να τηρούνται και τα τέσσερα κριτήρια. Αυτό θα δυσκολέψει πολλά κράτη, πιστεύω. Και ιδιαίτερα θα πρέπει να χαιρετήσουμε την ε, συμπερίληψη αυτού ασφαλείας ε, των ε, περιφερειών που βρίσκονται σε αυτό το phasing out με διατήρηση ενός ποσοστού από την χρηματοδότηση της προηγούμενης περίοδου. Ιδιαίτερα όμως θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις περιφέρειες οι οποίες ήδη τώρα βρίσκονται σε phasing out και πρέπει και αυτές να συμπεριληφθούν στο δίκτυο ασφαλείας. Επίσης, ένα ελάχιστο ποσοστό του 5% δαπανών ε, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να κατευθυνθούν στην ανάπτυξη, γιατί έχει αποδειχθεί ότι η πολιτική συνοχής, ε, η διαρθρωτική πολιτική θα πρέπει να ενισχύει την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Άρα λοιπόν θα πρέπει το 5% να απευθύνεται, να είναι ειδικά επιφυλαγμένο να προορίζεται ειδικά όχι για την ύπεθρο πλέον, αλλά για την ανάπτυξη στα αστικά κέντρα. Εν ελάχιστο 5%. Πρέπει επίσης να προχωρήσουμε πως γραφειοκρατικοποίηση προς απλούστευση των διαδικασιών, φυσικά με πάντα υψηλή σημασία των ελέγχων, αυτό είναι αναμφισβήτητο, τα διαρθρωτικά μέσα, τα μέσα του Ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να ελέγχεται πώς διατίθενται. Αλλά, αλλά για να μην γέμε και τα χλωρά μας με τα ξερά θα πρέπει να διαφυλάσσουμε την απαραίτητη λειτουργία, ευελιξία στη λειτουργία των δομών. Με ε, φυσικά αποδεδειγμένης ε, αξίας ελεκτικά μέσα τα οποία θα διαφυλαχθούν, αλλά όχι με υπερβολική ε, επιβάρυνση γραφειοκρατική και κόστος φυσικά που θα αναιρέσουν όλη την προσπάθεια. Και επίσης κλείνοντας ε, για να δώσω μια γεύση από τις θέσεις που εκφράζονται σε όλες, από όλες τις ομάδες στο Γερμανικό Κοινοβούλιο ότι η διπραγματεύση για τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο που συστήθηκαν ε, ήδη σήμερα μας ε, προβληματίζει όλους το γεγονό ότι υπάρχει λιγότερο, υπάρχουν μικρότερα ποσά για διανομή και γι' αυτό πρέπει πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε εάν χρειάζεται για τις περιφέρειες της μετάβασης που έχουν ένα ποσοστό ΑΕΠ από 75% περίπου σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο να ορίζεται ότι θα λαμβάνουν, και αυτό να είναι ο βασικός τη περιφερειακής μα πολιτική, ότι θα ε, λαμβάνουν λιγότερα κονδύλια, λιγότερη ενίσχυση. Εμείς ε, στη Γερμανία έχουμε βρει λύσεις αρκετά ικανοποιητικές και νομίζω ότι ο στόχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια συμπληρωματική μόνιμη κατηγορία για τις περιφέρειες μετάβασης πρέπει να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σακουράκης παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση και να εκφράσω την ε, δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι ο Επίτροπος έφυγε και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο. Θα Νομίζω ότι θα τον ωφελούσε αν άκουγε πολλά από όσα έχουν ε, ακουστεί εδώ. Ε, προκαταβολικά θα ήθελα να ενημερώσω τους ε, παραβρισκόμενους ε, για το γεγονός ότι και η Ελλάδα μέχρι το 2007 είχε πολύ ψηλούς ε, ρυθμούς ανάπτυξης. Θα θυμίσω στους περισσότερους ότι είχε ρυθμούς ανάπτυξης του 4,5%. Για να φτάσει όμως σήμερα αθρηστικά τα τελευταία τρία χρόνια να έχει ένα μείον του ΑΕΠ του 23% και ε, σε περίοδο ακόμα πριν την εκδήλωση της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά να σημειωθεί, όπως το αποδεικνύει και η πέμπτη έκθεση για την ε, πολιτική συνοχής, αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των ελληνικών περιφερειών και των ε, ελληνικών περιοχών. Τα λέω όλα αυτά τα πράγματα γιατί η πολιτική συνοχής για την οποία συζητάμε Κάθε άλλο παρά την συνοχή και την σύγκληση έχει προωθήσει, ε, διότι κατά την άποψή μας το κύριο ζήτημα που πρέπει κανείς να δει είναι πού κατευθύνονται και τι εξυπηρετούν τα κονδύλια τα Ταμεία Συνοχής και τα Περιφερειακά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη μου αποτελεί κοινό τόπο ότι οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αποτελεί κοινό τόπο ότι τα νέα κονδύλια όλο και περισσότερο θα υποτάσσονται όλο και περισσότερο στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, δηλαδή στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Βασικός στόχος του κεφαλαίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σήμερα, που υπηρετούν και οι κυβερνήσει των κρατών μελών φυσικά, είναι ένας. Να φορτώσουν τα βάρη της κρίσης στον λαό για να ανακάμψει η μονοπωλιακή κερδοφορία φτηνή, ακόμα πιο φτηνή εργατική δύναμη, μόνιμη αφαίρεση κατακτήσεων και δικαιωμάτων, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει τρόπος για τον καπιταλισμό να βγει από την κρίση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα κονδύλια κατευθύνονται σε έργα και δράσεις επιλέξιμες γιατί υπηρετούν αποκλειστικά την γεωφορία των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων. Δηλαδή υποδομές και δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, πράσινες τεχνολογίες κτλ. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Connecting Europe, όπου τα 10 δις για αυτό το πρόγραμμα αφαιρούνται από το Ταμείο Συνοχής και κανένας βεβαίως δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό τουλάχιστον σήμερα, ενώ στην ε, Επιτροπή της Ρέτζη είχαμε συζητήσεις. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι μειώνονται, ε, μειώνονται χρήματα, μειώνονται πόρα το Ταμείο Συνοχής όπως, όπως είναι το παράδειγμα της Ελλάδας Χθε ο Υπουργό μα είπε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 40% των χρημάτων αυτών. Στην ερώτησή μου από ποιου κινδυνεύει δεν μου απάντησε. Πιθανώ να μπορέσει κάποιο να μου δώσει μια απάντηση στο ζήτημα αυτό. Επομένω, ε, κατά την άποψή μου, είναι ψέμα ότι τα ταμεία συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούν την ανάπτυξη. Χρηματοδοτούν την κερδοφορία των ομίλων που αναλαμβάνουν τα έργα και τι πιο πολλέ φορέ έχουν και την εκμετάλλευσή του, όπω συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω και σε άλλε χώρε. Αυτό είναι το πρότυπο τη ανάπτυξη του που κατοστρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσει και τα κράτη-μέλη. Πού κατευθύνθηκαν όμω κυρίω τα χρήματα στην Ελλάδα, βασικά στι μεταφορέ και στι μεταφορικέ συνδέσει, όπου πρέπει να γνωρίζετε κατασκευάζονται ακόμα αυτοκινητόδρομοι για του οποίου εισπράττονται διόδια για κάποιου δρόμου οι οποίοι θα υπάρχουν στο μέλλον. Οι Έλληνε πληρώνουν από τώρα διόδια για δρόμου οι οποίοι δεν υπάρχουν, αλλά του καταβάλουν. Ε, Στι λεγόμενε ΣΔΙΤ η συμμετοχή των ιδιωτών φτάνει 8% και καμιά φορά είναι και μηδενική. Επίση, κατευθύνονται στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, όπου το τέλο για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια τα τελευταία τρία χρόνια αυξήθηκε κατά 8 φορέ ή σε, ε, στην επεξεργασία λιμάτων ή στη δημιουργία ερευνητικών κέντρων παρεξελών, όπω λέγονται, ερευνητικά κέντρα όμω τα οποία δεν συνδέονται με την ανάπτυξη και τι ανάγκε τη δόπια παραγωγή. Αυτές, όλα αυτά τα έργα ούτε θέσει εργασία εξασφαλίζουν και πολύ περισσότερο μόνιμες ή βιώσιμες ούτε παραγωγικές υποδομές που και με τα αστικά δεδομένα θα μπορούσαν κάπως να οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Γι' αυτό η Ελλάδα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, γι' αυτό η απόκληση είναι τόσο μεγάλη και σήμερα η Ελλάδα και άλλες χώρες απειλούνται να, να βρεθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο βγαίνει όμω ωφέλιμος από όλα αυτά τα έργα, όπω και τα στοιχεία δείχνουν το 40 με 45% των επενδύσεων στην Ελλάδα επιστρέφουν στη Γερμανία και όπω κάποιο ε, Επίσημο είχε σημειώσει. Στην Πορτογαλία αυτό φτάνει για ένα ευρώ που επενδύεται στην ε, ε, Πορτογαλία τα 85 λεπτά να επιστρέφουν στις χώρες οι οποίες είναι οι net contributors όπως λέγονται. Έτσι η ανάπτυξη για την οποία γίνεται λόγος είναι ανάπτυξη μόνο για μια, μεγάλη, για μια μερίδα των μεγάλων επιχειρήσεων η οποία όμως ταυτόχρονα θα συνοδεύεται από μια πολύ ανεμική ανάπτυξη γενικά των οικονομιών όπως ξέρουμε και ακόμα κι αν υπάρχει αυτή θα υπάρχει μια ε, εκτεταμένη και μόνιμη ανεργία που φυσικά δεν έχει τίποτα να κάνει με τις ανάγκες που ε, χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχή θα έπρεπε να κατευθύνεται σε έργα και υποδομές που πράγματι είναι ανάγκες και για τους, και για τους εργαζόμενους και για την ανάπτυξη όπως είναι αντιπλημμυρικά έργα παραδείγματο χάρη. Δεν υπάρχουν. Όπω είναι αντιπυρικά έργα. Δεν υπάρχουν. Όπω είναι ε, εκπαίδευση, σχολεία, όπω είναι υποδομέ, ε, όπω είναι παιδική σταθμή, ώστε να καλύπτονται και αυτέ τι τεράστιε ανάγκε που έχουμε στη χώρα μα, όπου αυτή τη στιγμή δεκάδε χιλιάδε παιδιά είναι εκτό παιδικών σταθμών, ή όπω είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι στα γεράματα δεν μπορούν να, να έχουν ούτε καν τα κέντρα εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων, τα οποία λόγω τη οικονομική κρίση και αυτά κλείνουν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε ότι εκφράζεται ένα το φάσμα απόψεων εδώ, από το τα πάντα πάνε στραβά στην Ευρώπη μέχρι το τα πάντα είναι υπέροχα στην Ευρώπη. Ε, ο κύριος Πατατάσκη, παρακαλώ, από την Βουλγαρία. Κατάρσκη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ, στην ευκαιρία αυτή της συνάντηση, για αυτό το κρίσιμο θέμα. Για την ε, μεγάλη αυτή συζήτηση για την πολιτική συνοχή, η οποία θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο που θα εγγυάται καλύτερη δημοσιονομική επιθαρχία αλλά και θα αποτελέσει εγγύηση μεταρρυθμίσεων σε αρκετούς κέρια σημασίας τομείς. Αυτό ασφαλώς θα συμβάλλει στην επίτευξη του κύριου στόχου μας, τη μείωση δηλαδή των αποκλήσεων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης και μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται είτε ως καθαρός εισφέροντα ή καθαρός εποφελούμενα του ευρωπαϊκού Πρέπει να αλλάξουμε θεώρηση. Τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα ευρωτικά ταμεία θα πρέπει να αξιοποιούνται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας εν όλο και την επιτάχυνση της σύγκλησης. Έτσι εποφελούνται τόσο τα καθαρό συσφέροντα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό όσο και τα καθαρός εποφελούμενα του ευρωπαϊκού προπολογισμού κράτη και εξασφαλίζεται η πιο αποδοτική ε, διάθεση των κονδυλίων. Για αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι η συζήτησή μας θα πρέπει να επικεντρώνεται σε αποτελέσματα και σε περιφέρειες. Θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε εταιρικέ σχέσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Οι επενδύσει στην ανάπτυξη τη υπαίθρου στην προκείμενη περίπτωση αποτελεί ένα, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα πρόοδου. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρώ το ενδεχόμενο, την ιδέα να προχωρήσουμε πιο μία ανάπτυξη των τοπικών ε, κοινωνιών, των περιφερειών με τη χρήση των εφορετικών ταμείων και προγραμμάτων από διαφορετικούς χώρους. Η ιδέα αξιοποίηση διαφόρων πόρων, ποικίλων πόρων, μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων ε, ποικίλων σε τοπικό επίπεδο και ταυτόχρονα στηρίξει την βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν είναι πολύ σημαντική για μας, πλην όμως προκειμένου να υλοποιηθούν όλοι οι στόχοι της ε, Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της πολιτικής συνοχής στην επερχόμενη περίοδο 2014-2020, εμείς στη Βουλγαρία φρονούμε ότι πρέπει να συντονίζονται καλύτερα τα ταμεία με ένα κοινό πλαίσιο, στρατηγικό πλαίσιο, και με ε, τις, συμφωνίες εταιρικής σχέσης αφετέρου. Και δεν ήθελα εδώ να σχολιάσω τον κανονισμό και κάποιες συγκεκριμένες πτυχές του, διότι πιστεύουμε ότι το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει καθαρές και εξαντλητικές πρόνοιες, διατάξεις, να εξασφαλίζει επαρκή ευελιξία για τα κράτη-μέλη, διότι πρέπει να μεριμνούμε εμείς για την κάλυψη των αναγκών σε περιφερειακό επίπεδο. Εμείς στη Βουλγαρία θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, αυτά τα ελάχιστο 2,5% επί του ΑΕΠ ως αρχή αναδιανομής. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις πιο φτωχές περιοχές. Με την αρχή αυτή δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πραγματική σύγκληση μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων και των περισσότερων ανεπτυγμένων περιφερειών. Χρειάζεται λοιπόν να στοχεύσουμε στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με την, με την αρχή που έχει προσδοριστεί για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και να βρούμε άλλες αρχές, σε παραδείγματι ΑΕΠ σε λόγο με την αγοραστική δύναμη ή κάποια άλλη ε, αρχή. Συμφωνούμε με τους θεματικούς στόχους για την προσοχή προγραμματική περίοδο. Δεν συμφωνούμε όμως ότι θα πρέπει να οριστεί ένα αποθεματικό 5% από το από τα ταμεία υπό το τρέχον στρατηγικό πλαίσιο διότι πιστεύουμε ότι το αποθεματικό αυτό δεν θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρηθούν οι αρχές της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου. Κατάλληλα συμφωνούμε με την θεματική συγκέντρωση, πρέπει να είναι πιο απτή η στόχη, δηλαδή η θεματολογία μάλλον είναι πιο απτή, αλλά χωρίς υπερβολικές ε, προϋποθέσεις οι οποίες ε, περιστέλουν την ε, δυνατότητα επιλογής, την ευελιξία δηλαδή από πλευρά των κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί χώρος για να εκφραστούν οι τοπικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες με προϋποθέσεις εξάντε, γιατί η εξάντε γιατι η εξαντε αριθμότητα για μας είναι πολύ σημαντική, την υποστηρίζουμε, θέλουμε, θεωρούμε δηλαδή ότι βοηθάει στην ε, υλοποίηση των στόχων, αλλά πρέπει να διαφυλαχθεί και η αρχή της αναλογικότητας, αναλογικότητας και αν σταματά σε ένα επίπεδο η ε, χρηματοδότης θα πρέπει να είμαστε θέση να παρακολουθούμε τους άξονες προτεραιότητας και να μην υπάρχει επιβάρυνση ως προς την... Ε, να μην εφαρμόζεται αυτή η επιβάρυνση για την περίοδο για την οποία ισχύει η άρση. Θα πρέπει να μας καθοδηγούν, πιστεύω, οι μακροοικονομικές προϋποθέσεις, μακροοικονομικοί όροι. Και να μην μιλούμε μόνο για δημοσιονομική πειθαρχία. Τα νέα δημοσιονομικά μέσα είναι καλά νομίζω. Για δε τις δαπάνες θα πρέπει πιστεύουμε να γίνει αποδεκτός ο ΦΠΑ για την ε, επερχόμενη προγραμματική περίοδο και τα τρέχοντα κριτήρια αποδοχής σε σχέση με το ΦΠΑ επίσης θα πρέπει να διατηρηθούν. Και τώρα προχωρώ σε επίπεδο χρηματοδότηση. Πιστεύουμε ότι λιγότερο ανεπτυγμένε περιφέρειε θα πρέπει να την χάνουν περισσότερε χρηματοδότηση, περισσότερε υποστήριξη. Δεν συμφωνούμε με την αρχή τη χρηματοδότηση του 75%. Υποστηρίζουμε την πρόταση για προκαταβολικέ πλήρωμέ από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ τα κράτη-μέλη, θεωρώντα πάντω ότι τα ποσά τα οποία προτείνονται είναι ανεπαρκή και δεν εξασφαλίζουν την ρευστότητα που χρειάζονται οι αρχές διαχείρισης. Εν τέλει, επιτρέψτε μου να σχολιάσω τα λόγια κάποιων άλλων συναδέλφων. Χρειάζεται, πιστεύουμε, στοχευμένη χρηματοδότηση στα κράτη-μέλη. Το δε κοινό στρατηγικό πλαίσιο δεν φαίνεται να ε, επιτρέπει την υλοποίηση του στόχου αυτού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διαρωτηθούμε ε, μήπως είναι προτιμότερο να οριστούν εθνικές αρχές, γιατί αυτές τους έχουν καλύτερα τη δυνατότητα και την ευελιξία για τη διαχείριση των σχεδίων. Και επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική γραφειοκρατία. η οποία οδηγεί σε φόβους και ανησυχίες και έτσι ίσως εξηγείται και το κακό ποσοστό απορρόφησης. Η θεματολογική συγκέντρωση λοιπόν περιορίζει την ευελιξία για τα κρατη Καθιστά πιο δυσχερή για τα κρατη την απευθεία στόχευση στις, ε, στους σπόρους και την ε, χρήση τους εκεί που χρειάζονται περισσότερο. Ευχαριστώ. Thank you very much uh, for this contribution from Bulgarian. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνεισφορά από τον εκπρόσωπο του Βαλγαρικού Κοινοβουλίου. Από ό,τι κατάλαβα είστε υπέρ για μακροοικονομική ερεσιμότητα. Ο επόμενος ομιλητής Ο κύριος Χρυσόγελος. Με συγχωρείτε για την προφορά του όνοματός σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήθελα να τονίσω ότι η συζήτηση που κάνουμε δεν αφορά μόνο τα θέματα των χρημάτων, αφορά την ουσία, το τι Ευρώπη θέλουμε, αφορά την κοινωνική συνοχή και αφορά προφανώς ε, και το θέμα της βιωσιμότητας. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα είναι βιώσιμη και γι' αυτό ε, είμαστε υπέρ της επικέντρωσης και στις ε, θεματικές προτεραιότητες, έτσι ώστε να ξέρουμε προς τα που διατίθεται οι δημόσια πόρη. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι πόροι, αλλά οι δημόσιοι πόροι πρέπει να επιτυγχάνουν την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα. Προφανώ χρειάζεται μεγαλύτερο προπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι για να επιτευχθεί αυτό και ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο, πρέπει να διασφαλιστούν ήδη πόροι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε πράγματι να μην εξαρτάται απόλυτα από τις συμμετοχές των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε όμως και αποτελεσματική χρήση των πόρων για να πετύχουμε τη σύγκληση πραγματικά και την κοινωνική συνοχή και την οικολογική βιωσιμότητα και κοινωνική βιωσιμότητα. Και γι' αυτό οι πολίτες και άλλοι μηχανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πόροι που διατίθενται δεν απορροφούνται απλώς, αλλά χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό για την κοινωνία, τους πολίτες, τη συνοχή και τη βιωσιμότητα τρόπο. Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου των περιφερειών αλλά και των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση των περιφερειακών σχεδίων τα οποία θα συμφωνηθούν μεταξύ του κράτους, του κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα στα αυτά που λέμε συμβάσει εταιρική σχέσης, τα partnership agreements, θα πρέπει να κατά τη δικιά μας πρόταση να περιληφθούν και οι περιφέρειες είναι συναποφασίζοντες και συνυπογράφοντες και να έχει διασφαλιστεί και ουσιαστική διαβούλευση. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό για να μιλάμε πραγματικά για περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή. Χρειάζεται όμως από την άλλη μεριά και η κάθε περιφέρεια, μια και είμαι και περιφερειακό σύμβουλος στη χώρα μου, στο Νότιο Αιγαίο, σε νησιωτικές περιοχές, χρειάζεται κάθε χώρα να διαμορφώσει ένα δικό της σχέδιο Κοινωνική συνοχή, γιατί μιλάμε για τη συνοχή και τη σύγκληση μεταξύ περιφερειών τη Ευρώπη, αλλά πολλέ φορέ παρόμοια σχέδια δεν υπάρχουν μέσα σε κάθε χώρα, μεταξύ των περιφερειών τη ίδια χώρα, αλλά ούτε καν στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας, γιατί σε μια αναπτυγμένη περιοχή, σε μια αναπτυγμένη περιφέρεια, υπάρχουν πολλέ φορέ περιοχέ που έχουν μεγάλη διαφορά κοινωνικών υποδομών, περιβαλλοντικών υποδομών, ανεργίας κλπ. Και τέλος, θα έλεγα ότι θα πρέπει κάθε χρηματοδότηση να συνεθεί με την ύπαρξη σχεδίων και ε, αποφάσεων για χωροταξικό σχεδιασμό, για να ξέρουμε δηλαδή τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται και τι μπορεί να γίνει σε κάθε περιφέρεια. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα υπολογιστεί η κατάταξη των περιφερειών στις τρεις κατηγορίες, δηλαδή αναπτυγμένη, ενδιάμεση κατηγορία και λιγότερο αναπτυγμένη, ε, θεωρούμε πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη στοιχεία τα οποία θα είναι και του 12, του 2012, έτσι ώστε πραγματικά να μπορούμε να μιλήσουμε για την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας που υπάρχει σήμερα, γιατί άλλα τα στοιχεία του 8 ή και του 9 και άλλα τα στοιχεία φυσικά του 12 και πολλές περιφέρειες μας έχουν παρουσιάσει και μελέτη εδώ στην Επιτροπή Επιστήμονας ότι ορισμένες περιφέρειες έχουν ήδη αλλάξει κατηγορίες με βάση τα στοιχεία του 2009 σκεφτείτε αν περιληφθούν και στοιχεία του 2012 με δεδομένο ότι σε πολλές, περι, χώρες, παράδειγμα στη δικιά μας, αλλά και περιφέρειες, το ΑΕΠ έχει πέσει κάτω από το 17-20-25%. Και βέβαια μελλοντικά πρέπει να επανεξετάσουμε το δίκτυο αυτό που είναι καθοριστικός για την κατάταξη των περιφερειών ή και των χωρών. Το ΑΕΠ δεν είναι ένας αντικειμενικός δείκτης, πρέπει να εισάγουμε και άλλους δείκτες περί βιασιμότητας, περί κοινωνικής συνοχή, για να μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για πραγματική εικόνα των περιφερειών και των χωρών. Ευχαριστώ πολύ. Ja, herzlichen Dank, Herr für diesen Beitrag. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσόγελο, για την παρέμβαση, για την ομιλία σας. Από Εθνικό τώρα Κοινοβούλιο, ο επόμενος ομιλητής, κύριος Χάμπης από την Ουγγαρία. Δεν τον βλέπω. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας, καλώς, να σας χαιρετήσω όλους ε, και να εκφράσω τη χαρά που σας βλέπω στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης μεταξύ βουλευτών Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συζητούμε την πολιτική συνοχή, συζητούμε τις, ε, εταιρικές, ε, τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης. Από πλευρά μου λοιπόν. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα σημείο, σε ένα θέμα, τον απλουστευμένο υπολογισμό. Γιατί είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει ο απλουστευμένος υπολογισμός να γίνεται σε εθνικό επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις των ε, ιδιαίτερων, των ειδικών κανονισμών των ειδικευμένων διατάξεων, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η εδαφικότητα κατά τρόπο πιο ευέλικτο σε ορισμένες περιπτώσεις και γι' αυτό θα θέλουμε να υποστηρίξουμε το 10% η δε πρόταση προτείνει για πέντε χρόνια ενιαία διαχείριση και μπορούν τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν μια πιο ευνοϊκή κατάσταση για τρία χρόνια. Για τη διαφάνεια και την απόδοση λογαριασμών με βάση τον κανονισμό. Θεωρούμε ότι οι προτινόμενες διατάξεις είναι ικανοποιητικές. Υποστηρίζουμε την πρόταση επίσης της εδαφικής ευελιξίας που μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω. Το τεχνικό πεδίο, το τεχνολογικό πεδίο εξελίσσεται ταχύτατα στην εποχή μας και γι' αυτό θεωρούμε ότι η τριετής προθεσμία για την διατήρηση της κατάστασης νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί. Οι προτάσει της Πολωνίας και τη Βουλγαρία για το θόρυβο θέμενης αξίας είναι πολύ ενδιαφέρουσες και όπως άλλωστε έχω πει και στο παρελθόν, ο φόρος προσθέμενης Αξία θα πρέπει και στο μέλλον να υπολογίζεται. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι για μας, και ιδιαίτερα από για την ιδιαίτερη μου πατρίδα, τη Βόρειο Ουγγαρία, Ε, έχουμε κίνδυνο εάν εισαχθούν πιο αυστηροί κανόνες για τις ε, περιφέρειες να αποκλειστούν και να περιοριστούν από ορισμένα μέτρα υποστήριξη οι ορισμένες κοινότητες της περιοχής μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση αυτή. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριος Τσέλλερ από τη Γερμανία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς, και εγώ θέλω να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου για την ευκαιρία αυτή της συνάντησης με τους εθνικούς βουλευτές. Είναι πολύ σημαντική η φάση στην οποία βρισκόμαστε. Πρέπει να ενισχύσουμε τις επαφές μας και να μην συναντιόμαστε μόνο μια φορά το χρόνο με τα open days. Τώρα ιδιαίτερα σε μια φάση όπου αναπτύσσονται οι συζητήσεις κατά τρόπο εντατικό. Ε, ιδιαίτερα ευγνωμόνιμαι προς τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων που έλαβαν το λόγο οι οποίοι υπεγράμμισαν τη σημασία της πολιτικής της διαρθρωτικής πολιτικής και μετά το 2014 και ότι τα το Διευθυντικό Ταμείο θα έχει μεγάλη σημασία για τις περιφέρειες, για την ανάπτυξη ιδιαίτερως ε, και, τη και τις θέσεις εργασίας. διότι δεν είναι δεδομένο, τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι θα συνεχιστεί η διαρθρωτική πολιτική μετά το 2014. Και γι' αυτό θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπή. Ε, Επίση, προ του συναδέλφου, παράκληση στα δικά σα, στα εθνικά κοινοβούλια, να αξιοποιείτε κάθε ευκαιρία που έχετε για να επηρεάσετε τις κυβερνήσεις σας και να τις καλείτε σε εθνικό επίπεδο να δείξουν περισσότερη κινητικότητα σε επίπεδο Συμβουλίου. Γιατί ακούμε και από τον εκπρόσωπο του, ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου ότι ναι μεν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέσει προτάσει, αλλά το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί, δεν ξέρουμε τι στάση θα τηρήσουν τα κράτη-μέλη στα ζητήματα που έχουν πλέον ανοίξει προ το μέλλον τη πολιτική συνοχή συνοχής, πολιτική πολιτικής το 2014. Ταυτόχρονα έχουμε ψηλού επίπεδου αξιωματούχου των κυβερνήσεων, οι οποίοι αμφισβητούν πολλές από τις ε, προτάσεις της περιφερειακής πολιτικής μέσα σε ένα πνεύμα λιτότητας στον προπολογισμό και φαίνεται να μην αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει η περιφερειακή πολιτική, η πολιτική για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Όταν τους καλούμε να εξηγήσουν ε, πώς θα δώσουν κίνητρα, δεν δίνουν απαντήσεις. Νομίζω ότι μέσω των διευθυντικών ταμείων, μέσω της ε, πολιτικής της συνοχής μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και στην ανάπτυξη και στην ε, απασχόληση. Ιδιαίτερα δεν θα ήθελα να αναφερθώ στον Γερμανό και μάλιστα Βαβαρό συνάδελφο, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολιτική, στη στρατηγική 2020 ως βάση της πολιτικής ε, συνοχής και ταυτόχρονα θα ήθελα να ζητήσω και εγώ στα διευθυντικά ταμεία να επικεντρωθούμε στην ύπεθρο, γιατί 70% των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν στα αστικά κέντρα, εκεί αναπτύσσεται η... Εκεί υπάρχει ανάπτυξη. Χάρη σε αυτά μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους στόχους Ευρώπης 2020. Έτσι λοιπόν, κοινωνική ενσωμάτωση, κατάρριψη των κοινωνικών αποκλεισμών, ανάπτυξη, κοινοτομία είναι στόχοι που μπορούν να εξυπηρετηθούν χάρη και στα αστικά κέντρα, γι' αυτό δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε ούτε τα αστικά κέντρα ούτε τα περιαστικά. Ο χώρος της υπαίθρου επεφολείται τα μάλα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, περίπου 40% στο πλαίσιο της όλης γεωργικής πολιτικής με τους πυλώνες υπαριθμών 1 και 2. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό, ότι υπάρχει από αλλού χρηματοδότηση. Λέμε. Ιδιαίτερα, δε, χαιρετίζω τις παρεμβάσεις εκείνες που μίλησαν για ενίσχυση, βελτίωση της ε, υπερσυνοριακής συνεργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει από πλευράς του τα κονδύλια για την υπερσυνοριακή συνεργασία να αναέρχονται στο 7% των μέσων για την πολιτική συνοχή και τη ερωτική πολιτική και να απλουστευτούν οι διαδικασίες για τη διάθεση των κονδυλίων αυτών σε περίπτωση περισσοριακής συνεργασίας, γιατί ακριβώς στις παραμεθορίους της ε, Ευρώπης, ε, μάλλον των κρατών μελών, ζει και αναπτύσσεται η Ευρώπη και αυτήν πρέπει να υποστηρίξουμε. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να και εκ μέρους ε, των προτάσεων που έχει διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση Περιφερειακής Συνεργασίας ότι χρειάζεται συνεργασία μέσα στην Ευρώπη αλλά και διεύρυνση της συνεργασίας ε, με τρίτα κράτη, κυρίως με τα κράτη της γειτονίας μας και αναζήτηση νέων μέσων όπως ε, μέσων γειτονίας ή προενταξιακών μέσων που μπορούν να αξιοποιηθούν στοχευμένα για να φέρουν καρπούς εκεί όπου χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσέλερ. Εκ μέρους της Επιτροπής. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Μάρτιν να λάβει το λόγο. Έχει, κάνει... Έχει πάρει πολλές σημειώσεις από τις παρεμβάσεις σας. Φαντάζομαι ότι σε κάποια θέματα να θέλει να δώσει πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Παρακαλώ. Thank you very much, Chair. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν εξαιρετικά πλούσια και ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση. Και ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι μπορούσαμε απευθείας να ακούσουμε και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων να εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα ανησυχιών. Φυσικά θα αναφέρουμε τα σχετικά στον Επίτροπο Χάν που δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο σύνολο της σημερινής συζήτησης. Άκουσα να εκφράζεται ευρία υποστήριξη για την πολιτική και για το επίπεδο της χρηματοδότησης που ο Επίτροπος Χάν είπε ότι πρέπει να παραμείνει, γιατί είναι μια πολύ σημαντική πολιτική, πολιτική συνοχή για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης μεγάλη σχέση με τα επιχειρήματα που ε, είναι απαραίτητα για να το πετύχουμε αυτό έχουν ε, και τα περί αποτελεσματικότητας της πολιτικής. Το έχουμε το στοιχείο αυτό συμπεριλάβει στην πρόταση της Κομισιόν ε, ώστε να δείξουμε ότι είναι αποτελεσματική πολιτική και πρέπει να γίνει και ακόμη περισσότερο. Δεύτερον, διασύνδεση με την στρατηγική Ευρώπη του 2020. Αναγνωρίζεται πλέον ευρέως ότι είναι πλήρως απαραίτητο και δικαιολογημένο να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση ενωσιακή πηγαίνει στις προτεραιότητες. Δεν είναι ασυμβίβαστη αυτή η στρατηγική, αλλά ευθυγραμμίζεται πλήρως με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν η ε, ανάγκη σε περιφερειακό επίπεδο και για να μπορεί η πολιτική συνοχή να εκπληρώσει τον ρόλο της μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης. Ετέθη το ζήτημα της θεματικής συγκέντρωσης. Ότι αυτό πρέπει να εξισορροπηθεί με την ευελιξία, δηλαδή οι περιφέρειες να μπορούν να καθορίζουν ε, τις δαπάνες, επειδή γνωρίζουν καλύτερα πού πρέπει να πάνε τα χρήματα. Ο Επίτροπος Χάν μίλησε σε εστίαση, στόχευση και σε ευελιξία. Δηλαδή πρέπει να ισορροπήσουμε τα δύο αυτά σκέλη. Όταν μιλάμε για συγκέντρωση, εννοούμε συγκέντρωση σε αρκετά υψηλά επίπεδα για επιθεματικών στόχων. Εάν δείτε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, η πρόταση τη Κομισιόν είναι η χρηματοδότηση να εστιαστεί σε τρει αρκετά ευρύ τομεί, δηλαδή έρευνα καινοτομία, στήριξη Ε και ενεργειακή απόδοση. Αυτό αφορά ένα ποσοστό τη χρηματοδότηση. 80% στι πιο ανεπτυγμένε, 50% στι λιγότερο ανεπτυγμένε. Επομένως, ουσιαστικά μιλάμε την, για την ευελιξία που την έχουμε συμπεριλάβει και έτσι μπορούν και οι περιφέρειες να αποφασίζουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια. Πρέπει όμως να δεχθούμε και τη διασύνδεση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Από πλευράς Κομισιόν, επειδή ο Επιτροπής χρησιμοποιεί αυτή την παρομοίωση με ένα μενού εστιατορίου. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει συμβατότητα με την προσέγγιση αυτή, δηλαδή να πούμε ότι από 11 πιάτα του μενού μπορούν τα κράτη να επιλέγουν 3 ή 4. Δηλαδή από τους 11 στόχους τους 3 ή 4 ε, στόχους να επιλέγουν. Και αυτό ενσωματώνεται στη γενικότερη προσέγγιση ότι δηλαδή πρέπει κάπως να προκαθορίζονται οι επιλογές για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Εν συντομία τώρα θα ήθελα να μιλήσω για τις συμβάσεις εταιρική σχέσης και την αρχή της εταιρική σχέσης. Το ουσιώδες στοιχείο της έννοιας μιας σύμβασης εταιρική σχέσης είναι συνδυασμό τη προσέγγιση από κάτω προ τα πάνω και από πάνω προ τα κάτω, αλλά όχι με μια άκαμπτη ε, προσέγγιση που θα ισχύει για όλε τι χώρε. Δεν νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε αλληλουχία, δηλαδή πρώτα να έχουμε τη σύμβαση και μετά να βλέπουμε τα προγράμματα. Θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο σχεδιασμός των προγραμμάτων και η εκπώνηση τη ε, σύμβαση εταιρική σχέση είναι κάτι που πρέπει να γίνει ταυτόχρονα. Θα ήταν πολύ θεωρητικό να ξεκινήσουμε δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο, στο επίπεδο κρατών και να φτάσουμε στα μεμονωμένα προγράμματα. Όχι, αυτό πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα από εκείνο διότι τελικά αυτή η συμφωνία ή Σύμβαση εταιρική σχέση αποτελεί μια αποκριστάλλωση αυτών που ε, αποτέλεσαν τα στοιχεία του σχεδιασμού του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα, πρώτα απ' όλα δεν είναι εφικτό να έχουμε διαπραγμάτευση επί μια σύμβαση εταιρική σχέση και όταν εγκριθεί αυτή να περνάμε στη συνέχεια στη διαπραγμάτευση των μεμονωμένων προγραμμάτων. Δηλαδή για πρακτικούς λόγους θεωρούμε ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια συνδυασμένη προσέγγιση. Μέσω τώρα της σύμβασης εταιρική σχέσης μπορούμε να δώσουμε ζωή στην αρχή της εταιρική σχέσης να παράσχουμε δηλαδή το μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα στους διαφόρους εταίρους ε, να εκπληρώσουν το ρόλο τους. Θα υπάρξουν κάποιες, κάποια διάκριση θα υπάρξει, δηλαδή θα δούμε πώς, ε, τι διευθετήσεις θα υπάρξουν. Επιλεγμένοι, αιρετοί εκπρόσωποι, περιφέρειες και άλλοι φορείς. Ο κώδικας συμπεριφορά, ο κώδικας διοντολογίας θεωρούμε ότι είναι μια καλή ιδέα γιατί δίνει ε, μια προσέγγιση. Ποιοι θα είναι οι ρόλοι που θα διανεμηθούν στους εταίρους. Και βέβαια ρόλος των εταίρων είναι ακριβώς να εξασφαλίσουν την νομιμοποίηση, την οικειοποίηση του προγράμματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις, την αιρεσιμότητα για να είναι αποτελεσματική πολιτική, είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις. Ξεφράστησαν επιφυλάξεις από εγώ νομίζω ότι οι εξάντε ερεσιμότητα, προϋποθέσεις δηλαδή που θα πρέπει να υπάρχουν ώστε να ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση θα πάει ε, ε, για τις σωστές δαπάνες. Είπαν κάποιοι ότι το σημαντικό είναι να μην τα καταστήσουμε όλα άκρος πολύπλοκα από την αρχή. Γιατί ο στόχος είναι να πετύχουμε οι επενδύσεις να εκπληρώσουν το σκοπό τους. Και αυτό το προσυπογράφουμε απόλυτα και ως Κομισιόν και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από τη δική μας πλευρά προς αυτήν την κατεύθυνση. Μακροοικονομική όρη, μακροοικονομική αρισιμότητα. Αρχικά υπήρξαν κάποιες έντονες επιφυλάξεις, αλλά νομίζω ότι όσο προχωράει η συζήτηση πλέον διαφαίνεται μια κατανόηση του ότι η πολιτική συνοχή δεν μπορεί να απομονωθεί από την οικονομική διακυβέρνηση και τις σχετικές ε, ρυθμίσεις οι οποίες συζητούνται και τίθενται σε εφαρμογή. Και εδώ νομίζω ότι το βασικό στοιχείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι δεν έχουμε στόχο σε καμία περίπτωση να τιμωρήσουμε κράτη-μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες. Στήριξη χρειάζονται αυτά τα κράτη, τα κράτη που έχουν υπερβολικό έλλειμμα. Αντιθέτως λοιπόν η πρόταση της Κομισιόν διατηρεί την ιδέα να υπάρχει μέγιστη κρατήση χρηματοδότηση για αυτές τις, ε, χρηματοδότηση για αυτές τις χώρες. Όταν όμως ένα κράτος μέλος δεν μπορέσει ε, αποτύχει να ακολουθήσει τις συστάσεις ε, στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης και αυτό συστηματικά, τότε μπαίνει σε εφαρμογή η αιρεσιμότητα. Δηλαδή θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη στήριξη στα κράτη-μέλη που τη χρειάζονται επειδή αντιμετωπίζουν οικονομικέ δυσκολίε, αλλά θέλουμε και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρχουν συνέπειε εάν τα κράτη-μέλη αποτύχουν να τηρήσουν τι συστάσει του Συμβουλίου. Αυτό νομίζω ότι καλύπτει τα βασικά ζητήματα. Και ολοκληρώνοντας θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα όλους και όλες για τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα που θέσατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάρτσιν έτσι ολοκληρώνεται η εκδήλωσή μας. Εκ μέρους της Προέδρου κυρίας Χιούμπνερ, σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ, για τη συμμετοχή σας, για τις πολύτιμες παρεμβάσεις. Εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάθαμε πολλά. Από, απευθείας από τις δικές σας παρεμβάσεις και αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό. γιατί είναι και η πρώτη φορά που συμμετέχει άμεσα στην ε, νομοθετική διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Συμμετέχουμε λοιπόν ισότιμα με το Συμβούλιο και έτσι όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Επιτύχαμε πιστεύω πολλά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φερρυπίν, εδαφική συνεργασία, όπου μας έχει πλησιάσει περισσότερο τι δικές μας θέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει φτάσει στο 3,5%, Εμεί θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το 7%. Αλλά θα ήθελα επίση να υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιδιώκει λύσει για μικρά-μικρά σχέδια, τα τετριμένα όπως τα λέγαμε, αλλά θέλουμε την διεκδίκηση αυτή και περισσότερη χρηματοδότηση να την συνδέσουμε για τις ε, παραμεθόρειες περιοχές, να τη διασυνδέσουμε με ε, πιο ευρείες δομές που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ε, δομές συνεργασίας και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε. Μια σειρά από θέματα ακούστηκαν σήμερα. Ο συνάδελφος από το Connecting Europe Facility για το δίκτυο ασφαλείας ε, υπογραμμίστηκε και μια ενδιάμεση κατηγορία που παρουσίασαν αρκετοί συνάδελφοι. Άρα δεν έχει ακόμα κριθεί αυτός ο αγώνας, είναι αμφίροπος. Θα δούμε βεβαίω και τι τάσει θα τηρήσει εν τέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά είναι πολλοί αυτοί μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι έχουν πολύ σαφεί ε, επιφυλάξει ω προ την ε, αυτή προσέγγιση τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νέε ιδέε που εκφράζονται από κάποιους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για την προαγωγή μιας ευρωζώνης, διαρθρωτική πολιτική, δηλαδή να υπάρχει ενίσχυση ειδικά για την ευρωζώνη. Τι θέτει ερώτημα βέβαια πώς θα το συνδυάσουμε αυτό, πώς θα το συνδέσουμε με τις μέχρι τώρα εφιστάμενες δομές, γιατί υπάρχουν ανάγκες για ολόκληρη την Ευρώπη, ορόσημο πρέπει να προσδιοριστούν όροι στήριξη στις πιο φτωχές ε, περιφέρειες, πιο αδύναμες περιφέρειες και δεν ξέρω πώς θα συνδεθεί αυτό με την νέα αυτή ιδέα της ε, ειδικής στήριξη για την Ευρωζώνη. Πρέπει και χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε προσωπικές μου προτιμήσεις λόγω της ε, ιδιαίτερης μου πατρίδας, πρέπει να δούμε πώς θα το συνδέσουμε. αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας και σας καλώ σε μια μικρή δεξίωση στο διάδρομο έξω από την αίθουσα. Ευχαριστώ και πάλι. Very good. So, now we have the cocktail. As it always is. You Yes, yes. A cocktail, yeah. Five minutes.